Colleagues, I can open the meeting um, again and... Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Συγγνώμη για όσους ήταν εδώ σε 9 το πρωί, καθυστερήσαμε λίγο. Θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση για τα όσα διαμήφθησαν στην συνεδρίαση των συντονιστών και φυσικά και τι ανακοινώσει του Προέδρου. Καταρχάς, για τους εισηγητές και τους συντάκτες γνωμοδοτήσεων, είχαμε δύο γνωμοδοτήσεις. Η μία, μία έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού για το 2010. Αυτή η κανονικά βάση του εκπεριτροπού συστήματος έπρεπε να πάει στους μη εγγεγραμμένους. Οι μη εγγεγραμμένοι δεν την ήθελαν και πήγαν στους επόμενους, δηλαδή στο ΕΛΚ. Θα καταρτήσουν λοιπόν μια γνωμοδότηση επί του θέματος αρμόδιος συντάκτης είναι ο κύριος Μαρινέσκου. Δεύτερη γνωμοδότηση για τους φιλελευθέρους, έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα κάνει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και επομένως η σύσταση των συντονιστών είναι εάν ε, ετοιμάσουν έκθεση από πλευρά Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, θα συντάξουμε και εμεί τη γνωμοδότηση. Αλλά αν δεν κάνουν έκθεση, δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε και εμεί γνωμοδότηση. Αυτή είναι η απόφαση λοιπόν. Δύο θέματα επιτροπολογίας. Το ένα, οι σαρωτέ ε, σώματος. Ε, συζητήσαμε για το ε, θέμα της επιτροπολογίας στο θέμα της ασφάλειας αεροπλοείας, ιδίως το θέμα της εισαγωγής των σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια και η πρόταση του Προέδρου ήταν να ληφθεί απόφαση μετά από τη διαβίβαση των ε, μέτρων. Ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι ακριβώς θα προτείνουν. Όταν θα λάβουμε την ενημέρωσή τους ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε και επί της διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε. Για τις άδειες των ε, κυβερνητών σκαφών αποφασίστηκε να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια πολιτική ομάδα που έχει αντίρρηση για τη διαδικασία για τις άδειες των πιλότων, να παρουσιάσει ε, σχέδιο ψηφίσματος. Ε, θα συζητηθεί αυτό στην συνεδρίαση των συντονιστών τον Αύγουστο και θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι παρούσα. Εάν κάποια λοιπόν από τις πολιτικές ομάδες έχει αντίρρηση για τη διαδικασία επιτροπολογίας για τις άδειες ε, των πιλότων, ε, μπορείτε να καταθέσετε σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο θα παρουσιάσουμε στους συντονιστές ε, στη συνεδρίαση του Αυγούστου. Είχαμε αρκετά θέματα στα διάφορα. Μία επιστολή δική μου για τις μελέτες που θα ζητήσουμε από το Τμήμα Πολιτικής για τον, από τον απομείνατο προπολογισμό του 2011 και επίσης κάποιες ενημερωτικές επιστολές στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία για την Ομάδα Εργασίας Προστασίας Δεδομένων, την οποία διαβιβάσαμε στην κυρία Λιχτεμπέργκερ και ε, για την, ε, το διάδρομο ανάπτυξης Βαλτικής Αδρατικής, ε, ε, με συνοδεία αρκετών αιτήσεων από τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου διαδρόμου. Υπήρχε και ένα αίτημα της ομάδας των Πρασίνων να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής της ε, έκθεση ίδια πρωτοβουλία του κυρίου Τέιλορ για τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά καμία από τι υπόλοιπε ομάδε δεν ήταν υπέρ τη επέκταση του πεδίου εφαρμογή και επομένω μένει ω έχει, κύριε Τέιλορ μόνο τα δικαιώματα των επιβατών ε, αεροπορικών πτήσεων και όχι όλων των μεταφορικών μέσων. Για το e-call ενημερωθήκαμε για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να είναι υποχρεωτική κότο η κόλε για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων οχημάτων μετά από το 2015, να γίνει μια πιο εκτεταμένη συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιες απόψεις για το τι θέλετε να συζητήσουμε, μπορείτε να το πείτε στους συντονιστό σας και να το συζητήσουμε στη συνεδρίαση του Αυγούστου. Η Ευρώπη των Συντηρητικών και Δημοκρατών ε, ζήτησαν ε, να εξετάσουμε ε, το θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων. Δεχτήκαμε την πρόταση γιατί υπάρχει περιθώριο για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, επομένως θα γίνει μια έκθεση επί του συγκεκριμένου θέματος και θα αποσταλούν και επιστολές ε, για τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ώστε να λάβουμε και την επίσημη έγκριση. Λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ε, εγκρίθηκε λοιπόν από πλευρά συντονιστών ε, η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια για τα προγράμματα χρηματοδότησης των υποδομών συμφωνήσαμε να καλέσουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μία από τις επόμενες συνεδράσεις προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη για τη δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων ε, υποδομών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα την πρώτη δέσμη ε, μέτρων για το σιδηροδρομικό πακέτο ε, αποφασίσαμε στους συντονιστές να επικεντρωθούμε στην αναδιατύπωση. Ε, διανεμήθηκε στους κοιόδης εισηγητές και στους ε, συντονιστές ένα σχετικό έγγραφο. Η εισηγήτρια, η κυρία Σερικιάνη, θα προσκληθεί στην συνεδρίαση των συντονιστών στις 30 Αυγούστου για να μας πει πώς έχει η κατάσταση για το θέμα αυτό. Μετά από αρκετές συνεδριάσεις με τους κοιόδης εισηγητές. να σας πω ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση ε, που έγινε σήμερα το πρωί ήταν ε, έγινε πολύ μεγαλύτερη πρόεδρος από ό,τι έγινε στα υπόλοιπα ε, συνεδριάσεις και ελπίζουμε η συγγήτρια να μας ενημερώσει στα τέλη Αυγούστου για το θέμα. Και τέλος, ε, οι πράσινοι ρώτησαν για το επίσημο αίτημα της Πολωνίας να μεταφερθούν 1,2 δις ευρώ από το προϋπολογισμό από το σιδηροδρόμου στα οδικά ζητήματα. Ε, εξετάσαμε με τη Γραμματεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί. Δεν υπήρχε τι επίσημο αίτημα της Πολωνίας για να γίνει η μεταφορά του κονδυλίου. Δεν υπήρχε λοιπόν επίσημη αίτηση από πλευράς Πολωνίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά λοιπόν για τα όσα διαμήφθησαν στην συνεδρίαση των συντονιστών. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ωραία, μπορούμε να εγκρίνουμε τα όσα σας είπα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Λογικά θα έπρεπε να είχαμε την ψήφιση της Σύμβασης των Αθηνών, αλλά αυτό αναβλήθηκε όπως γνωρίζετε για τον Οκτώβριο αν δεν κάνω λάθος. Επομένως στη συνέχεια έχουμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρασίνου Ακροτηρίου σχετικά με τις ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Ο Ντομινίκ Κρικέ είναι ο εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια οριζόντια, κλασική οριζόντια συμφωνία για τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πράσινο Κροτηρίου με στόχο να προσαρμοστούν διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν σήμερα, που έχουν συναυθεί μεταξύ πράσινων πρωτεύων και κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην κοινοτική νομοθεσία. Είναι λοιπόν, όπω είπα, μια κλασική συμφωνία. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η συμπερίληψη μιας ρήτρα ορισμού που αφορά όλες, ε, όλες τις μεταφορές υπάρχει δηλαδή ανεφόρον πρόσβαση στις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πράσινου Ακροτηρίου. Υπάρχει μια ρήτρα κατά των πρακτικών που στρέφονται κατά του ανταγωνισμού και επίσης ό,τι αφορά τη φορολόγηση του καυσίμου. Και αυτό αφορά τρίτες εταιρείες τρίτων χωρών που εκτελούν πτήσεις από προς Ευρωπαϊκή Ένωση Πράσινο Ακροτήριο. Είναι, όπως είπα, μια τυπική οριζόντια συμφωνία. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης. Πρέπει να δώσουμε την σύμφωνη γνώμη μας. Εγώ σας ε, συνιστώ να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της συμφωνίας, κύριε Πρόεδρε. Και εδώ ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ντομινίκ. Λέω ο Πρόεδρος, ο κύριος Αλκατράου, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε και σύμφωνα με τον εισηγητή. Πρόκειται για μια τυποποιημένη συμφωνία και για έναν από τους Ευρωπαίους εμπλεκόμενους που, θέλει, που επιθυμούν να έχουν, επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε σχέση με το πράσινο ακροτήριο και ανταποκρίνεται αυτό στη θέση μας η ομάδα μας μπορεί να ακολουθήσει την πρόταση του εισηγητή Συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο εισηγητής πρόκειται για μια τυπική, για μια κλασική συμφωνία σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των δημερών ε, συμφωνιών. Σε αυτή την οριζόντια συμφωνία συμφωνούμε με τη γραμμή του κύριου Ρικέ και πρέπει να τονίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα για όλες τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι θα απλουστευτεί η κατάσταση που χαρακτηριζόταν από ε, μεγάλη ποικιλομορφία διαφοροποίησης. Στηρίζουμε απόλυτα λοιπόν την πρόταση του κυρίου Πικέ και την έκθεσή του, του κυρίου Ρικέ, συγγνώμη. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Ρικέ και να πω ότι η ομάδα μας ECR θα στηρίξει τις γενικές γραμμές ε, της έκθεσής του. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρικέ για την έκθεσή του, αλλά και τα συμπεράσματα αυτής. Δηλαδή ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Είναι μια σημαντική συμφωνία γιατί πράγματι θα επιτρέψει να υπάρξει ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τις 8 διμερείς συμφωνίες. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της όλης εργασίας που εκπονούμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια. 47 τον αριθμό είναι οι οριζόντιες συμφωνίες που έχουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε βέβαια να διανύσουμε ακόμη αρκετό δρόμο. Θα το πράξουμε με τη δική σας βοήθεια και με αποφασιστικότητα. Ένα σχόλιο πέραν της ε, νομική συμμόρφωση αν θέλετε, αυτή η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία διότι πρόκειται για συμφωνία με μια χώρα που δεν είναι τόσο προηγμένη μεν, αλλά έχει μεγάλη ε, εξάρτηση από τον τουρισμό δε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή της. Η ανάπτυξη του τομέα των αεροπορικών μεταφορών είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό στοιχείο και η συμφωνία αυτή σίγουρα θα βελτιώσει την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή σας ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε για την έκθεση αυτή έχει ως εξής. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας το Σεπτέμβριο. Εν συνεχεία, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου ψηφίζουμε στην Ολομέλεια. Σεπτέμβριο, λοιπόν στην Επιτροπή μας και πρώτη σύνοδος του Οκτωβρίου. Τότε ψηφίζουμε επί της έκθεσης ΡΙΚΕ. Επόμενο σημείο, μέλλον του ΦΠΑ. Ανταλλαγή απόψεων. Με τον Μάρκους Φέρμπερ που είναι ο συντάκτης νομοδότης, δεν έχει έρθει ακόμη. Οπότε πρέπει λίγο να φλιαρίσουμε έτσι να περάσει η ώρα μέχρι να ε, έρθει ή καλύτερα να διακόψουμε. Καλύτερα να διακόψουμε κανένα δύο λεπτά μέχρι ότου φτάσει ο εισηγητής μας. Πότε προβλέπετε αυτό, γρήγορα φαντάζομαι. Λοιπόν, θα τον βρούμε, μην εξαφανιστείτε οι υπόλοιποι. Okay, colleagues, if we can restart. Μπορούμε να ξαναρχίσουμε. Έφτασε ο Μάρκους. Το μέλλον του ΦΠΑ λοιπόν. Μάρκους, γνωμοδότηση δική σου. Σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ζητώ φυσικά συγγνώμη διότι λόγω του χρονοδιαγράμματος όπως είχε δοθεί από τη γραμματεία ως Ευαγγέλιο της σημερινής συνεδρίασης βασίστηκα σε αυτό και γι' αυτό είχα και κάποια ανηλυμένη υποχρέωση, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να μην κατέστρεψα το πρόγραμμα των άλλων. Ε, να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το μέλλον του ΦΠΑ. Οδεί προς μια πιο απλή, πιο αποτελεσματική δυνατότητα συστημάτων ΦΠΑ. Πρόκειται για ένα πράσινο βιβλίο και όχι για κάποιες νομικές προτάσεις ε, για να το αναφέρουμε αυτό με σαφήνεια. Αλλά αυτό το πράσινο βιβλίο αναφέρει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που αφορούν το μέλλον του ΦΠΑ. Το, η πλειοψηφία των συστημάτων ΦΠΑ είναι πολύ περιπλόκα πράγματα. Έχουμε και όσον αφορά και τους ιδίους πόρους και την πρικοδότηση με ιδίους πόρους ένα πολύ ευάλωτο όσον αφορά πάτες ε, και παρατυπίες ε, σύστημα. Και γι' αυτό τα σημεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πράσινης βίβλου, του πράσινου βιβλίου, για μας για την Επιτροπή Μεταφορών είναι σημαντικό Πώς θα αντιμετωπίζετε το ΦΠΑ στον τομέα των μεταφορών. Διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο σε σχέση με την Ευρώπη είναι σημαντικό διασυνοριακά ανάλογα με τον φορέα των μεταφορών να έχουμε μια ξεχωριστή αντιμετώπιση του ΦΠΑ. Σε όλα τα κράτη οι ναυτιλιακές και εναέριες μεταφορές εξαιρούνται από το ΦΠΑ. Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία έχουν ειδικό καθεστώς για τους σιδηροδρόμους και τις πλωτές μεταφορές. Στη Γαλλία υπάρχει ένα σύστημα ΦΠΑ στο Εθνικό Σύστημα Ναυτιλιακών Πλωτών Μεταφορών. Στην Ελλάδα για τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, Πολωνία και Σλοβενία, ΦΠΑ για τη μεταφορά επιβατών οδικά. Και έτσι θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό το ευρύ φάσμα να το καλύψουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μορφές εξαιρέσεων. Εξαιρέσεις για άτομα όσον αφορά την μεταφορά τους ή για κάποια είδη αγαθών σε σχέση με τις μεταφορές και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε για να είμαστε πλήρεις. Στο πράσινο βιβλίο καταλήγει στο συμπέρασμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το ΦΠΑ ως τομέα στον τομέα μεταφορών είναι πολύ κατακαιρματισμένος ο τομέας αυτός και θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια να καταλήξουμε σε ένα ισότιμο δίκαιο πεδίο ε, εφαρμογής. Καταρχήν τρία πρότυπα μπορούμε να σκεφτούμε. Είτε όλα θα φορολογούνται είτε όλα δεν θα φορολογούνται. Αυτά είναι οι δύο απλούστερες, ας το πω προσεγγίσεις. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να προσέξετε. Σχεδόν δεν ακούσατε τα ότι έχω πει και θα μετά θέλετε να κάνετε αγαπητοί συνάδελφε εσείς ε, κάποια σχόλια. Ε, νομίζετε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε αλλά αυτό δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ουσιαστικά τρεις ε, θεμελιώδεις ε, δυνατότητες. Ξαναξεκινάω ώστε και τα λέω και πιο αργά για να τα καταλάβουν οι Αυστριακοί. Πρώτον, είτε πλήρως θα έχουμε απελευθέρωση από το ΦΠΑ ή δεύτερον, θα υπάρξει εισαγωγή πλήρους φορολόγησης με ΦΠΑ. Ή τρίτον, θα κάνουμε χρήση <clears throat> τέτοιων εξαιρέσεων ως γενικών κανόνων εφαρμογή. Δηλαδή, για όλους ε, τους ε, μεταφορείς πανευρωπαϊκά. Στη δική μου γνωμοδότηση που στα αγγλικά σας την υπέβαλα, διότι μια και πίεζε ο χρόνος δεν ήταν δυνατόν να έχουμε όλες τις μεταφράσεις στη διάθεσή μας έγκαιρα και για να έχουμε μια δυνατότητα να συνεννοηθούμε, και παρόλα αυτά να μπορούν να ασχοληθούν οι συνάδελφοι με το θέμα, γι' αυτό την κατέθεσα στα αγγλικά, επισημαίνω ότι αυτή τη στιγμή για την εσωτερική αγορά λόγω του κατακαιρματισμού του ΦΠΑ δεν έχουμε ένα έννοιο πλαίσιο. Έχουμε μια περίπλοκη και άδικη κατάσταση όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών και την ε, μεταφορά ε, σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών. Επισημαίνω ότι ο τομέας των μεταφορών όσον αφορά τη μείωση εκπομπών ρήπων μέχρι το 2050 θα έχει ειδικέ ευθύνε ε, και ε, καθήκοντα. Και αυτά όλα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη. Διότι ένας κατακαιρματισμένος τομέας ε, και ιδιαίτερα για το ΦΠΑ θα πρέπει να μας κάνει να πούμε ότι δεν είναι η πιο οικολογική προσέγγιση. Είναι μάλιστα και θα έλεγα η τάση προς την ε, αποφυγή των ευθυνών. Και εδώ ε, είμαι υπέρ του να υπάρξει η δυνατότητα χαμηλότερου ΦΠΑ ή μηδενικού ε, ΦΠΑ για κάποιες ε, περιπτώσεις και θα πρέπει σε σχέση με τις δυνατότητες αυτές από το, τον τόπο της εφαρμογής να έχουμε ενιαίες δυνατότητες εφαρμογής και να μην έχουμε εξαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών λόγω της πολυμορφίας των δυνατοτήτων ε, μεταφοράς πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή των βαρών όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Είναι το πιο απλό πρότυπο θα έλεγα αυτό και θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα άλλο πλαίσιο αυτή την αρχή εις φόρων προτείνει και γι' αυτό θα ήταν μια εφικτή δυνατότητα και στο πλαίσιο του ΦΠΑ μια τέτοια ρύθμιση να ε, εγκρίνουμε. Αυτά, εν πάση συντομία, αυτά που θέλω να προτείνω σε το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει στην αρμόδια επί της ουσίας ε, Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή να σεβαστούμε το δικό της χρονοδιάγραμμα. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί εκεί η ψηφοφορία προς έγκριση. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο εμείς πια αλλά ελπίζω ότι με την πρόταση που υπέβαλα, με βάση αυτήν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτό το στενό περιθώριο να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρκους. Χαίρομαι που δούλεψες γρήγορα και είχαμε το κείμενό σου στα αγγλικά γιατί έχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα και με την οικονομική και νομισματική. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι θα έχετε όλη την έκθεση στις γλώσσες σας μέχρι τις 22 Ιουλίου. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 23 Αυγούστου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί θα είναι καλοκαίρι, θα έχουμε διακοπές. Είπε και ο εισηγητής ποιο είναι το πρόβλημα. Έχει προχωρήσει γρήγορα η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ψηφίζει το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πάντως τον Μάρκους που και ο ίδιος προχώρησε ώστε τουλάχιστον να μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση. Ο κύριος ε, Καντρό για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στη... Θέλω να ευχαριστήσω σε σχέση με το συντάκτη γνωμοδότησης για αυτή την εισαγωγή και τις παρατηρήσεις του. Είναι ένα περιεκτικό σύντομο κείμενο, πλήρες ε, από την άλλη πλευρά, που αναφέρει την πολυσχηδή κατάσταση στα κράτη-μέλη και την ποικιλότητα που υπάρχει όσον αφορά τους διάφορους φορείς μεταφορών σε σχέση με το ΦΠΑ και οι διαφορές αυτές μεταξύ των επιμέρους φορέων στα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Αν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία κατάσταση πρέπει να εκπονήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται παντού σε όλα τα κράτη στις ίδιες αρχές. πιθανόν θα είναι δύσκολο, δυσχερές το εγχείρημα. Μια πλούστευση όμως είναι, είναι δεδομένο ότι πρέπει να επιτευχθεί και πρέπει να αναφερθεί και να προσθέσουμε πού το ΦΠΑ θα εισπράτεται, πού θα ε, επιβαρύνει μεταφορές και με ποιο τρόπο ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο. Η γραμμή αφετηρίας, η εκκίνηση να είναι δεδομένη σε σχέση με τον τόπο ε, κίνησης μιας ε, μεταφοράς και για, τον, για την ίσπραξη. Μια άλλη πτυχή είναι αποφυγή της, των απατών όσον αφορά το ΦΠΑ. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο τονίζεται στο πράσινο βιβλίο Υποστηρίζω τον συντάκτη γνωμοδότησης όταν λέει ότι είναι υπέρ σε ε, λιγότερες περιπτώσεις να υπάρχει ε, μηδενικό ή χαμηλό ποσοστό φορολόγησης με ΦΠΑ όταν πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες ε, όταν πρόκειται για περιβαλλοντικά κίνητρα που θέλουμε να δώσουμε οικονομικά κίνητρα που θέλουμε να ισχύουν. Η κατεύθυνση που ακολουθεί ο συντάκτης νομοδότησης νομίζω ότι είναι σωστή είναι σωστή η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός αυτός. Δεν βλέπω να υπάρχουν τριβές και συμφωνώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η κυρία Μέσνερ είναι η εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Ε, γνωρίζετε όμως ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να παρέμβει. Εξ ονόματός της λαπούμε λοιπόν ότι αυτή η έκθεση μας φαίνεται ενδιαφέρουσα, ακριβώς ε, λόγω των όσων μας είπε και ο εισηγητής, ε, λόγω της τρέβλωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το ΦΠΑ σε διάφορα ε, κράτη-μέλη. Κάποιες χώρες έχουν ΦΠΑ για τις εναέρειες μεταφορές και για τις θαλάσσιες μεταφορές, κάποιες άλλες όχι. Κατανοούμε λοιπόν ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το ζήτημα αυτό και επίσης ε, να εξετάσουμε και την ανάγκη εναρμόνισης με όλα τα μέσα μεταφορών. Επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο ο καθένας να πληρώνει το κατάλληλο τίμημα για τις μεταφορές. Δημιουργούνται όμως και άλλα προβλήματα για τον τρόπο υπολογισμού του ΦΠΑ. Πώ μπορούμε να υπολογίσουμε το ΦΠΑ κατά το τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικό και δίκαιο. Θα πρέπει να λαμβάνετε στην αρχή, θα πρέπει να λαμβάνετε στο τέλος. Τι γίνεται με τις ε, διεθνικέ μεταφορέ, ε, θα πρέπει να το σκεφτεί και αυτό ο εισηγητή. Θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση στο ΦΠΑ ή όχι. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ότι θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με εναρμονισμένες προτάσεις ε, και να έχουμε μια καλύτερη ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής αγοράς σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να αναλύσουμε καταλήλως τις προτάσεις του εισηγητού προκειμένου να μπορέσουμε να ε, έχουμε και συγκεκριμένες απόψεις στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Φέρμπερ για την έκθεσή του. Well, it's quite a complex issue and I'm certainly not the, the, the person that's an expert on Δεν είμαι βέβαια ειδική σε θέματα ΦΠΑ και φορολογίας εν γέννη, αλλά Σαφώς ε, είναι πολύ μεγάλο το φάσμα των συζητήσεων, το γνωρίζουμε και από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να δράσουμε και αυτό που υποστηρίζουμε είναι να μην αναλάβουν το βάρος του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις χωρίς λόγο ή να μην έχουν επιπλέον επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ. Το κόστος και η γραφειοκρατία θα πρέπει να ελεγχιστοποιηθεί για τις ε, επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές. οποιαδήποτε εξαίρεση θα πρέπει να περιοριστεί για να μην έχουμε κατακερματισμό. κατακαιρματισμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός λόγος να κάνουμε μια συζήτηση επί του θέματος, αλλά το θέμα, το θέμα είναι πώς θα προχωρήσει αυτό. Όσον αφορά τώρα τις αντιρρήσεις μας, εμείς είμαστε σαφείς και θεωρούμε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να έχουν άποψη επί του θέματος. Όσον αφορά τώρα τις μεταφορές, έχετε δίκιο. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες και κανονισμοί για το πώς ε, λειτουργούν οι μεταφορές και οι αγορές μεταφορών. Ο κύριος Φέρμπερ έκανε κάποιες προτάσεις στο σημείο 5 υποστηρίζει χαμηλότερη ή μηδενική ε, φορολόγηση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο μέσα μαζικής μεταφοράς. Εννοούμε μόνο τα λεωφορεία ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο διεξοδική η ανάλυση μας εδώ και επίσης υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Η χώρα καταγωγής, επί παραδείγματι. θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, διότι θα πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων ο τρόπος με τον οποίο ε, γίνονται οι χρεώσεις. Θα πρέπει να μας πει πώς θεωρεί ότι μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε λοιπόν κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις ε, για κάποια από τα σημεία που ανέφερε ο κύριος Φέρμπερ. Αυτά προς το παρόν. Όπως σας είπα, είναι περίπλοκη η συζήτηση, ιδίως στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Καλό θα ήταν όμως για τα σημεία που ενέφερα να μας διευκρινίσει λίγο περισσότερα στοιχεία ο εισηγητής και να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εξ ονόματος της ομάδας μας. Ο κύριος Κράμερ. Εγώ ευχαριστώ τον συντάκτη γνωμοδότησης για την έκθεσή του, για την γνωμοδότησή του. Πρέπει να πούμε ότι είναι άδικο μη κοινωνικό, μη οικολογικό αυτό που γίνεται στην Ευρώπη με το ΦΠΑ. Με οξυμένο τρόπο μπορεί κανείς να πει ότι οι τρόποι μεταφοράς που, δημιουργούν τη μεγαλύτερη ρήπανση, οι εναέρειες μεταφορές, επειδή στην στρατόσφαιρα απελευθερώνονται αυτοί οι ρήποι, απελευθερώνονται αυτές οι μεταφορές από το ΦΠΑ, οι άλλοι πληρώνουν και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και έχουμε 27 κράτη-μέλη, 27 25 έχουν σιδηροδρόμους και τα 25 πληρώνουν ΦΠΑ, ε, άλλοι όχι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η Ελλάδα μετά την κρίση 13%, η Γερμανία 19%, πρωτοπόρος. Αν από το Βερολίνο στις Βρυξέλλες πάμε το σιδηρόδρομο, όχι μόνο κρατάει τρεις φορές τόσο χρόνο η μεταφορά, αλλά τρεις φορές περισσότερο κοστίζει η επιβάρυνση όσον αφορά την φορολόγηση. πρέπει να γίνουν πιο φτηνά ε, τα εισιτήρια και έχουμε και την επιβάρυνση στο περιβάλλον αν δεν καλυφθούν οι ενέργειες μεταφορές, εκείνοι που ρηπαίνουν, αν ευνοούνται κιόλας ε, φορολογικά, είναι η λανθασμένη πορεία. Και ο, ο πολίτης, ο οποίος μία ή δύο φορές ε, παίρνει αεροπλάνο στη, κάθε χρόνο για να πάει κάπου, όμως ε, βλέπουμε ότι εκείνοι που πληρώνουν για 20 ταξίδια οι μάνατζερ, ε, όσοι εμπλέκονται σε επιχειρήσεις ε, ευνοούνται ιδιαίτερα και έχουν και φτηνότερα εισιτήρια και δωρεάν εισιτήρια γιατί οι απλοί πολίτες να επιβαρύνονται σε σχέση με τους άλλους που είναι τακτικοί ταξιδιώτες. Πρέπει να υπάρξει ένας εναρμονισμός και δεν μπορεί να είναι υπόθεση του κάθε κράτους μέλους. Πρέπει πανευρωπαϊκά να ρυθμίζονται τα πράγματα. Και ένα ακόμα πράγμα. Όταν μια ε, εταιρεία αερίων μεταφορών αγοράζει ένα αεροπλάνο δεν πληρώνει ΦΠΑ. Το ξέρατε, εγώ δεν το γνώριζα. Αν ένα σιδηρόδρομος ε, αγοράζει κάποια, ε, κάποιο κινητήρα, κάποιο τρένο, πληρώνουν ΦΠΑ. Ή κανένας δεν θα πληρώνει και δεν θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή όλοι θα πληρώνουν ΦΠΑ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εξαιρέσεις. Και στο 2, στο εδάφιο 2, περιγράφεται η κατάσταση σε σχέση με αυτή την αδικία. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να απαιτήσουμε ή όλοι θα πληρώνουν και θα επιβαρύνονται ή κανείς. Με το ίδιο δίκαιο πάντα, με την ίδια βάση, με την ίδια αρχή. Και δεν είναι δυνατό στη Γερμανία να έχουμε 19% και να έχουμε την πληρωμή εκεί που αγοράζει κανείς το εισιτήριο για παράδειγμα. Και το ίδιο σε σχέση με τις ε, εθνικές μεταφορές εκεί όπου αγοράζεται το εισιτήριο. Σε σχέση με τις σενάριες μεταφορές για παράδειγμα. Έχουμε μια ένωση μεταξύ Βερολίνου και Βραδενβούργου που 50 επιχειρήσεις συμμετέχουν εκεί και που κάνουν αυτή την, αυτόν τον επιμερισμό Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε με κάθε σαφήνεια, κάθετα, ότι απαιτούμε ή όλοι θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ ή κανείς και με τα ίδια ποσοστά, ώστε να υπάρχει ένα ενίο πλαίσιο και να είμαστε φιλοπεριβαλλοντικοί όσον αφορά τις μεταφορές. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα η έκθεση του εισηγητή και θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρέμβασή του. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να πω το εξής. Το θέμα του ΦΠΑ Πολλέ φορέ χρησιμοποιείται για να υπερφορολογικοποιήσουμε, αν θέλετε, τα πράγματα. Στην Πολωνία θελήσαμε να εισαγάγουμε το ΦΠΑ για τις λιμενικές υπηρεσίες, αναδρομικά μάλιστα, με αναδρομική ισχύ. Υπάρχουν ε, κάποιες πρωτοβουλίε, οι οποίε όμω δεν είναι σωστέ. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά στον τομέα των μεταφορών. Ο κύριος Φέρμπερ Κάνει λόγο επίσης για την ε, διαφοροποίηση των συντελεστών ΦΠΑ. Τι θέλει να μας πει ακριβώς, ότι πάντοτε θα πρέπει να έχουμε ένα μηδενικό συντελεστή ή πρέπει να υπάρχει απαλλαγή από το ΦΠΑ, γιατί δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, ε, τις δημόσιες συγκοινωνίες, μεταξύ αυτών. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά χρήζει περισσότερης διευκρίνησης. μέσω του ΦΠΑ θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφορών. Εσείς χρησιμοποιείτε και το οικολογικό επιχείρημα στην έκθεσή σας. Είναι σημαντικό μεν, αλλά υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα, υπάρχουν και άλλες πτυχές. Και υπάρχουν και καθαρά οικονομικού τύπου επιχειρήματα. Πρέπει, κατά την άποψή μου, να δώσουμε μια ευκαιρία και στους άλλους τρόπους μεταφορών μέσω των σιδηροδρόμων, των εσωτερικών πλωτών οδών. Επομένως νομίζω ότι καλό είναι να εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τον Ίση, γιατί εγώ προσωπικά θα το πράξω. Πάντως καλά κάναμε και θίξαμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριο Ρικέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω τον Μάρκο Φέρμπερ για την έκθεσή του που πραγματεύεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Τρεις μικρές παρατηρήσεις. Πρώτη, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων και εγώ φυσικά θα ήθελα να υπάρχει μια εναρμόνιση του ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε αρμονικά τα πράγματα. Βέβαια πρώτα απ' όλα μεταξύ των διαφόρων χωρών και μετά μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, όπως είπαν οι προλαλήσαντες συγκεκριμένα Λιμπεράτσκι και Κράμερ να χρησιμοποιηθεί το ΦΠΑ ως ένα αντισταθμιστικό εργαλείο ε, μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφορών. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η μοναδική μου από ό,τι φαίνεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δημόσιες συγκοινωνίες, ε, να ξέρουμε ότι κατά κανόνα επειδή είναι λιματικές επιδοτούνται οι δημόσιες συγκοινωνίες και δεν μπορούμε να μην έχουμε υπόψη μας ότι εισπράτεται ένα φόρο εντό εισαγωγικών για τι δημόσιε συγκοινωνίε. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε μια ισορροπία. Και το τρίτο σχόλιο μου, ουσιαστικά είναι μια πρόταση που θέλω να κάνω. Επειδή μιλάμε για το συντελεστή, για την εναρμόνιση του ΦΠΑ και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ΦΠΑ ως εργαλείο εναρμόνισης και ρύθμισης, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς αποδίδεται ή πού αποδίδεται ο ΦΠΑ. Έχουμε το δημοσιονομικό, το πολιετές πλαίσιο και έχουμε τους ίδιους πόρους τους ίδιους πόρους λοιπόν της Ευρώπης. Προτείνεται μια-δυο ποσοστές μονάδες του ΦΠΑ να ε, πηγαίνουν στους ίδιους πόρους. Μήπως θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε ε, ένα μέρος του ΦΠΑ για τις υποδομές, συγκεκριμένα ό,τι αφορά το ΦΠΑ για τις μεταφορές. Τώρα, αν δεν υπάρχει ΦΠΑ για την ε, αεροπορία, όπως είπε ο Μίκαλ Κράμερ, δεν ε, θα μπορεί εκεί ένα μέρος του ΦΠΑ να αποδοθεί σε αεροπορικές υποδομές, άρα εκεί η εναρμόνιση δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια πρόταση και να πούμε ότι ένα, μια ποσοστία μονάδα ΦΠΑ, κάποιο, κάποια μονάδα θα μπορούσε να αποδοθεί για τις υποδομές. Αυτό είναι χρήσιμο. Και όχι μέσω της επιστροφής στο γενικό προϋπολογισμό. Νομίζω για τις μεταφορές θα ήταν πιο χρήσιμο να υπάρχει ίσπραξη και μετά διανομή, κατανομή του ποσού στις διάφορους τρόπους μεταφοράς. Νομίζω αυτό θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ραπώνη από την Κομισιόν έχει το λόγο. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή λοιπόν παρουσίασε στην Πράσινη Βίβλο. Στόχος της ήταν να ξεκινήσει η συζήτηση. Η φορολογία, ο ΦΠΑ για ε, το, για του τρόπου μεταφορά και τη χρήση των μέσων μεταφορών είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν συντάξει ένα ειδικό δελτίο. Είναι σωστή ανάλυση του εισηγητή. Η διαπίστωση είναι ότι η σημερινή κατάσταση είναι αρκετά πολυσχεδής και τερόκλητη σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και την αντιμετώπιση του ΦΠΑ ε, στους διάφορους τρόπους μεταφορών. Διαφέρει η κατάσταση από το ένα κράτο μέλος στο άλλο και αυτό οδήγησε σε ένα είδος στρέβλωση του ανταγωνισμού και ε, σε μια πολύπλοκη εφαρμογή του καθεστώτος ΦΠΑ και κατακαιρματισμό της αγοράς. Εξού και η Κομισιόν θα ήθελε να δοθεί μια αρκετά ξεκάθαρη απάντηση από πλευρά των φορών εκμετάλλευση του Κοινοβουλίου των κρατών μελών για να δούμε ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι προφανέ όμω ότι σε αυτό το στάδιο η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να παραμείνει ω έχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ε, είτε είναι για οικονομικούς, για οικονομικούς, για περιβαλλοντικούς λόγους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και θέλουμε να υπάρξει μια σαφής θέση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον ε, τον τομέα των μεταφορών. Η Κομισιόν βάσει των δημόσιων διαβουλεύσεων προτίθεται το 2013-2014 να ε, δημοσιεύσει και μία πρόταση οδηγίας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε ε, Φέρμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Επειδή όλοι εξέφρασαν ότι δεν είναι ίσονο σημασία σε αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και το θέμα του ΦΠΑ είναι κάπως πιο περίπλοκο. Δεν ήθελα να τα πω όλα εξαντλητικά. Συνάδελφε Κράμερ, το γεγονό ότι μια επιχείρηση δεν πληρώνει ΦΠΑ, αυτό δεν σημαίνει προτέρημα αυτόματα. Ακούστε τουλάχιστον μία φορά συνάδελφε, προσέξτε. Ήθελα να σας πω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά τα ξέρετε φαίνεται όλα. Και επειδή σε σχέση με την ε, ε, ευνοϊκότερη μεταχείριση φορολογικά θα πρέπει να δει ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους δυνατότητα. Και πρόκειται για το θέμα προ, ε, εισφορά στην πηγή ή όχι. Και σε σχέση με την επιβολή του ΦΠΑ, όταν υπάρχει ε, επιστροφή, όταν υπάρχει δυνατότητα ίσπραξης στην πηγή, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής επειδή έχουμε το πρόβλημα των συγκοινωνούντων των, των δοχείων και όταν έχουμε ένα, ε, το πρόβλημα του ΦΠΑ για μια επιχείρηση δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό επειδή έχουμε αυτά τα δοχεία που επικοινωνούν. Εγώ λέω ότι όλα θα πρέπει να επιβάλλονται με ΦΠΑ. Και γι' αυτό αυτό το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος Λιμπεράσχη υπάρχει διαφορά μεταξύ μηδενικού ΦΠΑ και μη υποχρέωσης ε, καταβολής ΦΠΑ εγώ προτείνω όλα να είναι υπόχρεα προς καταβολή ΦΠΑ, αλλά να υπάρχει μειωμένο συντελεστής ΦΠΑ ή να πλησιάζουμε για κάποιες χρήσεις και το μηδενικό ποσοστό ΦΠΑ από πλευράς προσέγγιση. Εγώ λέω για τις δημόσιες μεταφορές να έχουμε ξεχωριστή αντιμετώπιση. Είμαι πρόθυμος να το συζητήσουμε συνάδελφε. Δεν ξέρω αν σε σχέση με το πράσινο βιβλίο για τον ΦΠΑ ή για τον καθορισμό των δημόσιων κρατικών μεταφορών αν θα το κάνουμε αυτό σε σχέση με στοιχεία που έχουμε για παράδειγμα για τις ε, κοντινές ε, αποστάσεις ε, στις δημόσιες μεταφορές να δούμε πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί όταν θέλουμε να καθορίσουμε τι ακριβώς είναι δημόσια, δημόσιες μεταφορές γνωρίζοντας ότι δεν είναι απλό θέμα ο ορισμός και ο προσδιορισμός γενικά για τις, ε, την ίσπραξη ΦΠΑ, γενικά πρέπει να δούμε πού θα υπάρχει υποχρέωση ίσπραξης καταβολής ΦΠΑ. Θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στη δεκαετία του 1990, τότε με τον Επίτροπο Μόντι, είχε επισημάνει ότι κάποτε θα εφαρμοζόταν η αρχή της χώρας προέλευσης. Δηλαδή στο σημείο προέλευσης ή εκκίνησης, εκκίνησης ενός ταξιδίου ή εκκίνησης μεταφοράς αγαθών ή στην αγορά ε, Εμπόρεύματο στον τόπο αγοράς εμπορεύματο θα πρέπει να εισπράτεται. Διότι όλο το σύστημα απατών απορρέει από το ότι δεν έχουμε την αρχή του, της χώρας ε, εκκίνησης αλλά, ε, η χώρας προέλευσης αλλά την χώρα στην οποία καταλήγει το εμπόρευμα ή η μεταφορά. Και γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις απατών. Γι' αυτό λέω πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως η αρχή της χώρας προέλευσης και να το δούμε αυτό στον τομέα μεταφορών. Θα πρέπει να είναι ο γενικός κανόνας αυτός για να μειώσουμε τις περιπτώσεις απατών. Αυτόματα θα μειωθούν με αυτόν τον τρόπο. Και άλλα σημεία σε σχέση με αυτό τα οποία ε, καλύπτω και αναφέρω είναι, αν δείτε τις προτάσεις για τον φόρο συναλλαγών, το τέλος ε, επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με τις ε, χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πάλι ως ιδέα δεν είναι τα χρηματιστήρια να χρησιμοποιηθούν, αλλά ο τόπος της χρηματοοικονομικής συναλλαγής. Εκεί να εισπράτεται το τέλος αυτό, ο φόρος αυτός. Ένα είδος αρχής χώρας προέλευσης ή τόπου προέλευσης για την ίσπραξη αυτή. Πρέπει να πω ότι γενικά έτσι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα με την εφαρμογή της χώρας προέλευσης ή χώρας εκκίνησης. Ο κύριος Κατράου είχε θίξει το θέμα σε σχέση με την ίσπραξη και η κυρία Μπιλμπάου επίσης. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Η δική μου πρόταση είναι, επειδή ως θέμα αρχής το θεωρώ σωστό όσον αφορά το ΦΠΑ συνολικά, είναι η, χώρα της, η αρχή της χώρας προέλευσης. Θα χαιρόμουν αν με ακολουθούσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής, διότι απλουστεύει αυτή η αρχή τα πράγματα. Αυτό θέλουμε, να απλουστευτούν τα πράγματα, να γίνουν ασφαλέστερα τα πλαίσια για την αντιμετώπιση απατών και πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη. Κύριε Ρικέ, ένα θέμα το οποίο καλύψατε είναι ένα ευρύτατο θέμα όσον αφορά την δέσμευση των φόρων, την χρήση των φόρων για συγκεκριμένες χρήσεις για τον τομέα μεταφορών σε σχέση με το ΦΠΑ για παράδειγμα. Δεν έχουμε τίποτα για την χρήση ε, πόρων ε, και είχαμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να αφήσουμε αυτόν τον τομέα και όσον αφορά και την Ευρωβινιέτα και ε, συνάδελφε Ερκαντράου, ξέρετε για ποιο πράγμα κάνω λόγο εδώ έτσι δεν είναι όμως στο ΦΠΑ που είναι διαφορετικό δηλαδή ένας γενικός φόρος, μια ίσπραξη γενικού τύπου φόρου που εισπράτεται, για να το δεσμεύσουμε, να δεσμεύσουμε αυτό το πόρο για συγκεκριμένη χρήση, θα είχα προβλήματα εγώ να το δεχτώ. Αν έχετε εσεί τροπολογίε που θέλετε να διατυπώσετε, να καταθέσετε, να το ξανασυζητήσουμε. Διότι στο τέλο τέλο θα έχουμε δημόσιου προπολογισμού που θα είναι δεσμευμένα τα κονδύλια για συγκεκριμένε χρήσει καθοριστικά και πρέπει να το δούμε αυτό αν δικαιολογείται από τα κράτη-μέλη να υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις. Είναι όμως ε, θέμα χρήσης ε, πόρων ή χρήσης κονδυλίων και έτσι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ και χαίρομαι για τις τροπολογίες που θα καταθέσετε και αμέσως μετά τις θερινές διακοπές Πρόεδρε θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα και θα το ξαναδούμε ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φέρμπερ. Να σας τα ξαναπώ, μετάφραση σε όλες τις γλώσσες του σχεδίου γνωμοδότησης μετά από τις 22 Ιουλίου θα τις λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 23 Αυγούστου 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Και ενημερωτικά η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπής, θα ψηφίσει στις 19 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας και καλωσορίζω τον κύριο Πάτρικ Κάλτιν, τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας τον κύριο Φρανκ Τερίνγκς από το ICAT ε, για θέματα ασφαλείας, Διευθυντή Πολιτικής ε, Αεροπορίας του Βελγίου και η κυρία Πατρίσια Ρεβέρδη είναι εδώ, η οποία είναι απληρώτια Γενική Γραμματέας, υπεύθυνη προγραμμάτων ασφαλείας. Θα θυμάστε, συνάδελφοι, ότι η Επιτροπή μας αποφάσισε να προσκαλέσει την ΑΕΚΑΤ να παρουσιάσει τα προγράμματά της, ιδίως τα θέματα της ασφάλειας, της αεροπορίας και της τεχνολογίας και την αξιολόγηση των ε, ε, σαρωτών υγρών και σαρωτών ασφαλείας. Αυτό ακολουθεί την φασαρία που είχαμε στα τέλη Απριλίου φέτος όσον αφορά τις ε, τη λήξη της ε, απαγόρευσης της μεταφοράς υγρών ε, για τους επιβάτες και ανησυχία που υπάρχει ότι θα μπορούσε να υπάρξει και ανάλογη αναταροχή το 2013 όταν θα εκπνεύσει και η προθεσμία για την ε, απαγόρευση των υγρών. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν να έρθει εδώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και αν μου επιτρέπετε να σας το πω αυτό, ε, καταλήξαμε σε απογοήτευση διότι τα μέλη ε, της Επιτροπής μας λαμβάνουν διάφορα μηνύματα από ε, διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και το μήνυμα που λάβαμε από όλους είναι ότι ποτέ κανείς δεν μας είπε κάτι ε, για το οποίο να συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι. Οι κατασκευαστές των μηχανημάτων μας λένε ότι τα μηχανήματα είναι έτοιμα. Κάποιες χώρες Ιδίως η Γαλλία λένε ότι τα μηχανήματα δεν είναι έτοιμα και υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που λένε ότι τα μηχανήματα είναι στη διάθεσή τους, ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που δέχτηκαν, ε, με τα χαράς δέχτηκαν τη χρήση των μηχανημάτων. Το θέμα ήταν ότι εμείς εδώ ως Κοινοβούλιο δεν ξέραμε ποιος μας λέει την αλήθεια. Έτσι προήλθε και η ιδέα της ανταλλαγής απόψεων με την υπηρεσία σας. Σας καλωσορίζω. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει πρώτος το λόγο. Λογικά θα πρέπει να έχετε λάβει όλη και την παρουσίαση. Θα υπάρξει και μια παρουσίαση επί της οθόνης. Δεν ξέρω ποιος θα αρχίσει. Εσείς θα αποφασίσετε. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσω εγώ. Λέγομαι Πάτρικ Καντήλ, είμαι αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής ε, Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας. Μάλλον και του, Γαλλικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα ως ΕΔΠΑ να σας παρουσιάσουμε σήμερα τις απόψεις μας και να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης θα ήθελα να σας εκφράσω τις, ε, τη λύπη του Προέδρου μας, κυρίου Ράντου, ο οποίος θα ήθελε να είναι εδώ, αλλά είναι σε αποστολή στη Σιγκαπούρη και δεν μπόρεσε για πρακτικούς λόγους να είναι εδώ σήμερα αλλά αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη συνάντηση αυτή, εξού και το γεγονός ότι συνοδεύομαι από τον Φραγκ Ντιουρέγκ ε, που είναι από το Βέλγιο, από το εστιακό σημείο του Βέλγιου για την ασφάλεια και ο οποίος ουσιαστικά θα κάνει τη σημαντικότερο τμήμα της παρέμβασης, της παρουσίασής μας. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν το έργο της ΕΔΠΑ σε θέματα ασφάλειας και κυρίως ό,τι αφορά την τεχνολογία, τεχνολογικά θέματα. Ελπίζω αυτό να είναι η επαρχή ενός οικοδομητικού διαλόγου, γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή, πράγματι έχουν υπάρξει παρανοήσεις και ασάφειες. Η παρουσίασή μας λοιπόν ξεκινάμε κάποια λόγια πρώτα απ' όλα για το τι είναι ΕΔΠΑ, Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά θα σας περιγράψουμε τις δραστηριότητες μας ε, στον τομέα της ασφάλειας και συγκεκριμένα σε σχέση με τα υγρά, αλλά και ε, του αρωτές σώματος. Εν τέλει θα κάνουμε κάποιες προτάσεις, ε, θα προβούμε σε κάποια καταληκτικά συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν ιδρύθηκε το 1955 και είναι ένας από τους περιφερειακούς οργανισμούς ε, που θα έλεγα έχουν από τους πιο σημαντικούς που έχουν ιδρυθεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΕΣΕΗ. Στόχος είναι η εναρμόνιση κάποιων κανόνων και μέτρων σε θέματα αεροπλοείας. 44 είναι τα κράτη-μέλη της ΕΔΠΑ. Στόχος μας είναι η ασφάλεια της ε, αεροπλοείας, η ασφάλεια και διευκόλυνση των επιβατών και το περιβάλλον. σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πολιτικής ε, αεροπορίας. Η κατευθύνσει της ΕΘΠΑ στον τομέα της ε, πολιτικής ασφάλειας ορίζονται με ένα έγγραφο αναφοράς που είναι το έγγραφο 30, DOC 30. Είναι ένα πρωτοποριακό έγγραφο, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και πρέπει να σας πω ότι αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι προσανατολισμοί κατευθύνσεις βασίζονταν σε αυτό το έγγραφο, το DOC 30. Ένα έγγραφο το οποίο καθορίζει αναλυτικά στοιχεία για διάφορα θέματα. Και σήμερα ε, είναι συμβατό με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους το έγγραφο αυτό, το οποίο έχει και παραρτήματα τα οποία ε, περιλαμβάνουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική ασφάλειας. Επίσης, ε, προτείνεται πρακτική βοήθεια στα κράτη-μέλη και αυτό χάρη σε ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Πρώτα απ' όλα τους ελέγχους ασφάλειας της ΕΔΠΑ. Παρέχουμε επίσης βοήθεια σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και ανάπτυξη εκπόνησης εγγράφων εργασίας, εσωτερικών εγγράφων εργασία για κάθε χώρα. Τέλος, έχουμε μια κοινή διαδικασία αξιολόγησης ε, ε, του εξοπλισμού ασφαλείας. Νομίζω ότι σχεδόν τα μισά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα παροχής βοήθειας από την ΕΦΠΑ και αυτό βέβαια ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο μέσα σε αυτή την περίμετρο των 44 κρατών μελών. Είμαστε οργανωμένοι σε δίκτυα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το δίκτυο των Γενικών Διευθυντών στο κρατών μελών. Είμαστε η ανώτερη εξωματικοί στις χώρες μας και έχουμε ευθύνη και αρμοδιότητα για τις χώρες μας σε θέματα ασφάλειας, της αεροπορίας και έχουμε και αρμοδιότητες ρυθμιστικού χαρακτήρα. Οι εμπειρογνώμονές μας συμμετέχουν στην ειδική ομάδα εργασίας, στην Task Force της ΕΔΠΑΛΑ και σε υποομάδες οι οποίες εκπονούν το σύνολο των τεχνικών κανόνων και προτύπων. Έχουμε επίσης έναν τρόπο εργασίας ο οποίος βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην διαβούλευση, στη συνεννόηση με τους αερομεταφορείς, τα αεροδρόμια, τους κατασκευαστές εξοπλισμού και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης συνεργαζόμαστε πολύ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μάλιστα σχεδόν πάντοτε παρίσταται στις ε, συνεδριάσεις μας και τη λαμβάνουμε πολύ υπόψη και έχουμε και ε, συναντήσεις ε, με τη Διευθυντική Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, τη ΔΟΠΑ και με την, Αραβική διάσκεψη πολιτικής αεροπορίας. Έχουμε και διμερείς επαφές όμως με μη ευρωπαϊκά κράτη όπως είναι η Σιγκαπούρη όπου ακριβώς βρίσκεται ο πρόεδρός μας σήμερα ή ε, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να προωθήσουμε και επίση κοινέ γραμμέ για την ασφάλιση αεροπορίας σε διάφορες χώρες του κόσμου. Θα δώσω τώρα τον λόγο στο φίλο μου Φρανκ Ντουρένξ, ο οποίος θα σα παρουσιάσει το πιο αναλυτικό τεχνικό μέρος της παρουσίασής Ευχαριστώ Πάτρικ. Συνεχίζω με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΚΑΚ. Το πρόγραμμα εργασίας ΕΚΑΚ προετοιμάζεται, εγκρίνεται και εφαρμόζεται σε τριετής κύκλους για την ασφάλεια. Τόνισα εδώ κάποια από τα κύρια στοιχεία του τρέχοντος προγράμματος ως εξής το μείζον μέρος ε, του προγράμματος εργασίας είναι υποστήριξη της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας στα κράτη-μέλη. Συν ε, επιπλέον δράσεων κατάρτισης ε, και εφαρμογής. Εδώ σε αυτό το πεδίο έχουμε και προγράμματα ελέγχου audit programs στα κράτη-μέλη της ίκα και με τις ύπα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η, ΚΑΚΑ δραστηριοποιείται έντονα στα προγράμματα αρρωγής ε, με βάση τα επιμέρους κράτη, συμπληρωματικά, παραπληρωματικά στο έργο της ε, ε, Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων και έχουμε μία προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο όσον αφορά την ασφάλεια στις ενέργειες μεταφορές νέες απειλές και αντίμετρα. Για παράδειγμα, κυβερνοτρομοκράτες, ε, δυνατότητες υιοθέτηση μέτρων αποτροπής. Επιπλέον, η προσέγγιση μας λαμβάνει υπόψη μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων, αξιολόγησης ε, ευάλωτου χαρακτήρα και ε, δυνατότητα να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μέτρα αποτροπής. Επιπλέον στο πρόγραμμα εργασίας μας, ειδικά όσον αφορά τον εξοπλισμό για την ασφάλεια, η έχει εκπονήσει τεχνικές προδιαγραφές και κοινέ μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τις ασκήσεις και δοκιμές υπό κοινή αιγίδα, κοινή αξιολόγηση εξοπλισμού ασφάλειας, η CEP. Περισσότερα γι' αυτό υστερότερα στην παρουσίασή μου. Συνεργασία με άλλες περιοχές του κόσμου που τονίζεται ως θέμα στο πρόγραμμα εργασίας, η υποστηρίζει περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως περιφερειακά σεμινάρια, θεματολογικά για θέματα ενδιαφέροντος. Επίσης δυνατότητα οικοδόμησης ε, δυναμικού ώστε να υπάρχει δυναμικό σε σχέση με τα κράτη-μέλη, διάχυση πληροφοριών και των πρακτικών όσον αφορά θέματα όπως τον έλεγχο της ποιότητας, συνεργασία με τα κράτη-μέλη που έχει κυριαρχικό πρωταρχικό ε, ε, ρόλο. Για τις τεχνικές και τεχνολογικές προδιαγραφές έχουμε την Task Force ICAC που είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο φόρουμ επαϊόντων όσον αφορά θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε αυτή τη συνεισφορά αυτή τη Task Force για τι προτάσει που υποβάλλονται από πλευρά τη για τι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς. Έχουμε ε, τα θέματα όσον αφορά τεχνική και προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και κοινέ μεθόδους δοκιμασιών που εφαρμόζονται από τα διαφορετικά δοκιμαστικά κέντρα για να διαπιστωθεί αν ένας εξοπλισμός, συγκεκριμένος εξοπλισμός ανταποκρίνεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή όχι. Και έτσι περιγράφονται τα είδη εκρηκτικών που πρέπει να μπορούμε να ανοιχνεύουμε με τις συσκευές μας. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το εγχείρημα. Αν ε, δείτε ότι χρειάζεται η έγκριση 44 κρατών ε, όταν έχουμε εθνικές, ε, εθνικούς καταλόγους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη που τονίζονται από αυτούς τους καταλόγους συγκεκριμένα θέματα περισσότερο έναντι κάποιων άλλων. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να πετύχουμε συνενετικό πλαίσιο εφαρμογής μέχρι σήμερα. Θεωρούμε ότι η διαβούλευση με τους διαφορετικούς τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας είναι θεμελιώδους σημασίας. Έχουμε καθορίσει μηχανισμούς για να επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. Για παράδειγμα, ε, συνεδριάσεις ε, για την πληροφόρηση όσον αφορά τους παραγωγούς τέτοιου εξοπλισμού για κοινέ διαδικασίες αξιολόγησης ή παραγωγοί προσκαλούνται να κάνουν παρουσιάσεις σε αυτή την Technical Task Force για τα όσα ε, εκπονούν και σχεδιάζουν. Επίσης έχουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη τα οποία δεν ανήκουν στην ΙΚΑΚ όπως Αυστραλία και Ισραήλ ώστε να υπάρξει όφελος για αυτά τα θέματα από αυτή τη συνεργασία και να προωθηθούν οι διεθνείς προδιαγραφές που θα υιοθετηθούν για την κοινή διαδικασία αξιολόγηση, αξιολόγησης, η κοινή διαδικασία αξιολόγησης εξοπλισμού που προανέφερα. Εν συντομία βασίζεται σε μια συμφωνία μεταξύ 43 των κρατών μελών μας να διαχέουν πληροφορίες και στοιχεία όσον αφορά τις δοκιμασίες εξοπλισμού ένα εγχειρίδιο τυποποιημένο έχει εκπονηθεί καθορίζοντας τις τυποποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζονται, ο ρόλος κάθε ενός που συμμετέχει και οι μέθοδοι όσον αφορά ανείχνευση εκρηκτικών ε, ανείχνευση υγρών εκρηκτικών και σαρωτές ασφάλειας. Δοκιμασίες γίνονται αιτήσια και συμμετέχουμε σε δοκιμαστικά κέντρα τα οποία καθορίζονται από τις εθνικές αρχές με την τελευταία προσθήκη σαρωτών ασφάλειας που θα αρχίσουν τις δοκιμές τους εφέτος. Οι εκθέσεις γνωστοποιούνται στα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν τα κράτη-μέλη τις αναγκαίες πληροφορίες για να πιστοποιείται ο εξοπλισμός ή να μην πιστοποιείται ανάλογα με την κρίση των κρατών μελών. Μια κύρια αρχή είναι η διαφάνεια. Εξοπλισμοί που ανταποκρίνονται σε σχέση με αυτές τις προδιαγραφές δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Και έτσι τα όσα αναφέρονται ε, σε σχέση με αυτά τα θέματα ε, ε, είναι προσπελάσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα στον ιστοτόπο. Είναι μοναδική στην Ευρώπη αυτή η δομή. Δίνουν, δίνει πληροφορίες στα κράτη-μέλη ώστε επικουρικά να βοηθήσουμε στην πιστοποίηση. Αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο βασίζεται στην προθυμία κάποιων κρατών μελών που έχουν εθνικό δυναμικό δοκιμασιών ώστε από κοινού να συνεργάζονται προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας. Λειτουργεί αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο και θα πρέπει να όταν έχουμε συμφωνήσει επί ενός καταλόγου οι τεχνικές προδιαγραφές ακολουθούν, συμφωνούμε για τις διαδικασίες, γίνονται οι έλεγχοι και συντάσσονται εκθέσεις απλές διαδικασίες με πολύ σημαντικά αποτελέσματα και συντονισμό που διασφαλίζει την επιτυχία. Αυτή η διαδικασία επέτρεψε τους ρυθμιστές και τη βιομηχανία να αναγνωρίσουν τους περιορισμούς και τα όρια της τρέχουσας τεχνολογίας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτοί οι περιορισμοί και θα χρειαστεί χρόνος και επενδύσεις από τις βιομηχανίες για να υποστηριχθεί περαιτέρω έρευνα και να προχωρήσουμε παραπέρα για την ε, σάρωση τώρα υγρών, αεροσόλ και γέλης. Αυτό το τμήμα αφορά την ε, εξέταση των υγρών, αεροσόλ και γέλης. Σάρωση και απαιτήσει βρίσκουμε τις, τους κινδύνους και τον τρόπο ανταπόκρισης. Το πλαίσιο και η συγκυρία όλοι θα θυμόσαστε ότι η απειλή αυτή εντοπίστηκε το 2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά, όταν υπήρχαν κάποια σχέδια τρομοκρατών να καταστρέψουν αεροπλάνα με υγρά εκρηκτικά τα οποία οι συναθουργοί θα ε, οδηγούσαν στο να εκραγούν στα ε, αεροπλάνα. Ε, τα υφιστάμενα μέτρα για την ασφάλεια και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν σε θέση να ανοιχνεύσουν αυτά τα υγρά εκρηκτικά και ιδιαίτερα δεν μπορούσαν να διαφοροποιήσουν αυτά τα υγρά από απλά κοινά υγρά. Η άμεση αντίδραση η απουσία τεχνικής λύσης ήταν ο περιορισμός της μεταφοράς υγρών, αεροσών, αεροσό και ε, γέλης παράλληλα άρχισε έργο για να καθοριστεί ο τρόπος αποτροπής και αντίδρασης ώστε να μπορούν να επιτρέπονται υγρά υπό την προϋπόθεση ελέγχων. Ελέγχων με την προϋπόθεση των όσων θα είχε καθορίσει η Task Force και τα όσα θα ίσχυαν από τεχνικούς κανονισμούς. Η Task Force υιοθέτησε και εκπώνησε μέθοδο για συστήματα ανείχνευσης τέτοιων υγρών πιλωτικά έγιναν δοκιμές το 2009 για αυτές τις μεθόδους. Το Δεκέμβριο 2009 ο Γενικός Διευθυντής της ε, ΙΚΑΚΑ συμφώνησε να ε, θεσπιστεί ένα πρόγραμμα από πλευράς ε, της ΙΚΑΚ για την αξιολόγηση εξοπλισμού ασφάλειας και να ξεκινήσουν δοκιμές, δοκιμασίες. Ήταν το δεύτερο πρόγραμμα αυτό. Μετά εκείνο το οποίο υφίστατο όσον αφορά συστήματα ανείχνευσης εκρηκτικών σε σχέση με τον εξοπλισμό και την επίδοσή τους για δοκιμές, δοκιμασίες, έχουμε τέσσερις τύπους ε, χαρακτηριστικά ανάλογα με τις δράσεις. Τύπος Α, ανείχνευση υγρών. Απαιτείται όμως να είναι ανοιχτό ε, το κουτί ή ε, το δοχείο. Τύπος Β, παραμένουν οι σφραγίδες σε κλειστό το δοχείο Τρίτον, διαφορετικά δοχεία ταυτόχρονα ξεχωριστά από την μεταφερόμενη ε, αποσκευή. Και τέταρτον, μέσα στην μεταφερόμενη αποσκευή στο αεροπλάνο. Έχουμε προγράμματα ελέγχων ακολουθώντας μια κοινή μεθοδολογία ελέγχων εφαρμόζοντας ε, στα τρία ε, κέντρα δοκιμών στην Ελβετία, την, το Κέντρο Αστυνομίας με το Fraunhofer Institut στη Γερμανία και το Ίδρυμα TNO στην Ολλανδία. Οι εκθέσεις για αυτές τις δοκιμές και δοκιμασίες γνωστοποιούνται στις αρχές των κρατών μελών της ΙΚΑΚ. Εν περιλήψη στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ιστοτόπο της ε, ΙΚΑΚ, στην ιστοσελίδα μας. Για τις επιδόσεις όσον αφορά τις δοκιμασίες δοκιμές τύπου α, β, γ και δ από το Μάιο 2010 έχουν μετατραπεί. Έχουμε δύο συλλογικές ε, τέτοιες ε, ε, δοκιμές α, β, γ τον Αύγουστο 2010, Ιανουάριο 2011. Πάμπολα συστήματα δοκιμάστηκαν. Μια τρίτη εκστρατεία βρίσκεται υπό εξέλιξη που θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του έτους η δυνατότητα εξέβρεσης, ανείχνευσης όσον αφορά τις μεταφερόμενες από τους επιβάτες ε, αποσκευές στο αεροπλάνο ε, βρίσκεται υπό εξέλιξη. Όσον αφορά τις ε, δοκιμές ε, όσον αφορά τους τύπους ε, α, β, γ και την ανταπόκρισή τους σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτός ο κατάλογος ε, αντιστοίχησης θα πρέπει να μπορεί να διευρύνεται σε σχέση με περαιτέρω δοκιμασίες και τεστ. Η παραγωγή διαρκώς βελτιώνουν τις επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρότι χρειάζεται χρόνο αυτή η ανάπτυξη, ο εξοπλισμός πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να μπορούν τα υγρά ε, εκρηκτικά να ε, ανοιχνεύονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θέματα εφαρμογής, υλοποίησης, σάρωση υγρών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς ε, λειτουργίας αεροδρομίων, προσδοκίες σε σχέση με τους επιβάτες, απαιτήσει ρυθμιστικών αρχών και μέσα στους περιορισμούς από πλευράς αεροδρομίων θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα αεροδρόμια με τέτοιου είδου ε, σαρωτέ, πρέπει να λαμβάνονται αποφάσει ε, για τον τύπο που θα χρησιμοποιείται να αγοράζουν και να χρηματοδοτούν την αγορά αυτών των ε, στοιχείων, αυτών των μηχανισμών και να μπορέσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τυποποιημένες διατάξεις και να υπάρξει η κατάρτιση των υπαλλήλων που θα χρησιμοποιούν αυτούς τους σαρωτές. Επίσης οι ε, επιβάτες πρέπει πλήρως να είναι ενημερωμένοι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους δοκιμασίες με σαρωτές. Οι αβεβαιότητες ε, σε σχέση με τα όσα θα ισχύουν σε σχέση με διαφορετικά αεροδρόμια ή διάφορους ε, προορισμούς θα είναι εις βάρος των επιβατών. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ε, αβεβαιότητες. Θα πρέπει να διευκολύνονται οι επιβάτες ε, και να γνωρίζουν τι θα συμβαίνει καθώς επίσης και να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με τα εγκεκριμένα υγρά. Λαμβάνοντας υπόψη το τι θα γίνεται σε σχέση με το σχεδιασμό τέτοιου είδους κέντρων οι ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κεντροποιημένα τέτοια, μονάδε, τέτοιες μονάδες. Ε, ένα, ένας για παράδειγμα Σαρωτήσα ανα πτέρυγα αεροδρομίου θα πρέπει για ένα συγκεκριμένο αριθμό δρομολογίων αεροπλάνων ή ε, διαδρομών να χρησιμοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Οι εταιρείε εναέριων μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα τους τύπους α, β, γ και δ απαιτώντας ε, να ε, ελέγχονται ξεχωριστά τα δοχεία μεταφοράς υγρών. Τα αεροδρόμια θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τις ανεφαντικημένου, ε, την ανεφαντικημένου ενεργοποίηση συναγερμών και το τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τον εξοπλισμό τύπου Δέλτα, που είναι ο εξοπλισμός που αναμένουν όλοι για να μπορέσει να λειτουργήσει, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αναμένουν να μπορεί να ανοιχνεύει αποσκευέ που μεταφέρονται στο αεροπλάνο και για ε, στερεά εκρηκτικά και άλλα. Όσον αφορά βιομηχανικές πτυχές, ο παραγωγός θα επικεντρώνει σίγουρα την προσοχή του στην βελτίωση της ανείχνευσης και της μείωσης των άνευ συναγερμών, ιδιαίτερα για τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τύπων και συστημάτων σε σχέση με τους χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα υγρά και τα, σύστημα, τα συστήματα ΔΕΛΤΑ και ε θα πρέπει να αναμένεται ότι όσον αφορά την δυνατότητα ανείχνευσης στερεών ε, εκρηκτικών ε, να βελτιώσουν τα πράγματα. Έτσι θα βελτιωθεί το δυναμικό ανείχνευσης και για τα στερεά και για τα υγρά εκρηκτικά αποφεύγοντας το ποσοστό ανεφαντικημένου συναγερμών και μειώνοντας το σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Η παραγωγή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες όσον αφορά την πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την προθεσμία του 2013. Κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει από πλευρά τη ότι θα μειώνεται η απειλή και θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και ότι τα δοχεία μεταφοράς ε, υγρών θα ε, ελέγχονται αποτελεσματικά. Πρέπει να αναπτύσσεται και να εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες αυτές θα είναι συμβατές με τα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όσα ισχύουν στα επιμέρους κράτη-μέλη. Αν οι διαδικασίες αυτές ε, δεν θα προβλέπουν σημαντική μείωση του κινδύνου, τότε αυστηρότερα μέτρα θα μπορούν να εφαρμοστούν και να εγκριθούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου στο εθνικό επίπεδο ώστε να προστατευτούν οι πολίτες. Τώρα, Ποιε είναι οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στοχεύουμε με επιτυχία να αντιμετωπίσουμε την προθεσμία του 2013 που έχει καθοριστεί από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τότε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν σαρωτικέ μεθόδου αποτελεσματικά. Πολλέ προκλήσει πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι λύσει θα πρέπει να υποπτεύονται ο κατάλογος θα πρέπει να είναι το δυνατόν ευρύτερος για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η ΕΚΑΚ θα εντείνει τις προσπάθειές της καθώς όλο και περισσότερο θα έχουμε τις δυνατότητες ε, δοκιμών. Τα αεροδρόμια που εποπτεύονται από τις εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν προγράμματα εφαρμογής και, σχέδια τα οποία θα προσαρμόζονται για τις ανα... ανάγκες λειτουργίας των αεροδρομίων θα πρέπει να υπάρχει διευρωπαϊκός συντονισμός για την επόπτευση της ε, ετοιμότητας και για την διασφάλιση ότι αυτή η σάρωση και αυτή η ανείχνευση θα διασφαλίστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέματα που ταυτοποιούνται σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει με συντονισμό να αντιμετωπίζονται πριν από την εκνοή της προθεσμίας του 2013. Διεθνής συντονισμός παγκόσμια απαιτείται για να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα ασφάλειας θα εναρμονιστούν ή θα είναι συμβατά μεταξύ τους και να αποφύγουμε διαφορετικά μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται ανάλογα με τον κάθε ξεχωριστό προορισμό. Το επόμενο μας θέμα είναι σαρωτές ασφάλειας η υλοποίηση της ε, μεθόδου των ε, ανιχνευτών των σαρωτών ασφάλειας ε, <clears throat> σε μια διαφορετική φάση οδήγησε την ΙΚΑΚ να δραστηριοποιηθεί για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να ισχύουν και θα βοηθήσει η ΙΚΑΚ αναφερόμαστε στα βήματα προς την ανάπτυξη αυτών των στοιχείων και σκιαγραφώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και ταυτοποιώντας και εντοπίζοντας τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επιτυχή εφαρμογή που είναι η αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων. Με απλά λόγια, η στόχη τη της άρρωσης επιβατών είναι να διασφαλιστεί ότι ο ένας επιβάτης ή ο άλλος δεν θα μπορεί να αποφύγει, να υπεκφύγει έλεγχο. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τον, ε, την ψηλάφιση ή τον ε, έλεγχο ε, μέσω προσωπικού ασφαλείας. Οι σαρωτές ασφάλειας οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνολογίες και δυνατότητα ανείχνευσης οποιασδήποτε ανομαλίας και ουσιών ή στοιχείων πέρα από τα ρούχα του επιβάτη, ιδιαίτερα τα μεταλλικά αντικείμενα. Το 2008 η Task Force για τα τεχνικά θέματα της ΙΚΑΚ ανέπτυξε τέτοιου είδους προδιαγραφές και απαιτήσει για τους αρωτές ασφάλειας, για την ανείχνευση διαφορετικών κατηγοριών αντικειμένων. Μια παρόμοια προσέγγιση όπως αυτή που περιγράψαμε προηγούμενα για τα υγρά έχοντας έτσι καθορίσει τον πίνακα απειλών, τον κατάλογο απειλών, μία μέθοδος μεθοδολογικά αναπτύχθηκε και ε, υιοθετήθηκε από πλευράς Γενικού Διευθυντή το Δεκέμβριο 2008 και επιπρόσθετα τα κράτη-μέλη τα οποία δοκιμαστικά κάναν, ε, κάναν τέτοιες δοκιμές ε, σαρωτών ασφάλειας στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρήχαν και συνεχίζουν, συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες για θέματα τεχνολογικής προόδου και <clears throat> μια ανταλλαγή πληροφοριών με την Αρχή Ασφάλειας των Μεταφορών των ΗΠΑ διασφαλίζει την ε, συμβατότητα στην αντιμετώπιση διατλαντικά των θεμάτων αυτών όσον αφορά τους ε, διατλαντικούς ε, διαδρόμους. Είμαστε έτοιμοι σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος σαρωτών και είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές. Συνεργαστήκαμε πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ΙΚΑΚ και με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της, ε, ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για μια επιτυχή αντιμετώπιση των σαρωτών ασφάλειας όταν θα δοθεί άδεια λειτουργίας τους, καθώς και με έναν κατάλογο όσον αφορά των συμβατών αυτών σαρωτών, έχοντας εκπονήσει τις αρχές προσέγγισης και εφαρμογής με τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα αεροδρόμια, κατάτηση υπαλλήλων και το εξίσου σημαντικό ενημέρωση πληροφόρηση επιβατών. Καλοχαιρετίζουμε την υιοθέτηση των νέων κανονισμών από την ε, Ρυθμιστική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα που είναι ένα κέρια σημασίας βήμα προς τα εμπρός Επίσης ενθαρρύνουμε έντονα τους, ε, παρα, τους, ε, τις εταιρείες που ε, παράγουν τέτοιου είδους εξοπλισμούς να προβούν στην εκπόνηση μηχανισμών ανείχνευσης απειλών, ανάλυσης στοιχείων κινδύνου και επισήμανση άμεσα στους όσους είναι υπεύθυνοι για αυτές τις συσκευές, για αυτές τις συσκευές ανομαλιών που διαπιστώνονται. Ολοκληρώνω, πρωτού περάσουμε στο γύρο ερωτήσεων-απαντήσεων. Θέλω να ε, τονίσω τα εξή στοιχεία που εμπνέουν την προσέγγιση της ΣΥΚΑ όσον αφορά την ασφάλεια σε νερείς μεταφορέ. Πρέπει να πετύχουμε ένα πλαίσιο αποτελεσματικότητας για την ασφάλεια όσον αφορά και τις προσδοκίες των επιβατών. Η μεταβατική περίοδος που χρειάζεται προς ένα νέο πρότυπο, συνδυάζοντας προδιαγραφέ και πρότυπα για την ασφάλεια, οδηγώντας τη βελτίωση δυνατοτήτων όσον αφορά τους ελέγχους επιβατών σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ας μάθουμε, ας συναγάγουμε μαθήματα από τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, οδηγώντας σε ένα ενιαίο πλαίσιο, διασφαλίζοντας ότι θα αντιμετωπιστούν ε, οι κίνδυνοι με τις προσδοκίες που θα έχουμε. Πρέπει να βασιστούμε σε μια ανάλυση κινδύνου για να αντιμετωπιστούν οι απειλές καθώς επίσης και νέων τεχνολογιών που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα και ανάπτυξη ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τρίτον, πρέπει να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες που θα διασφαλίζει σημαντικά τους επιβάτες στο κοινό και τις αξίες της κοινωνίας μας. Αυτά πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών μας. Η πρόθεση της εμπιστοσύνης, οι ευρωπαϊκές αξίες δεν είναι κάτι το δεδομένο. Αφορούν ακριβώς τον πυρήνα της ίδιας της Ευρώπης. Μαθήματα από όλες τις περιφέρειες και περιοχές δείχνουν ότι πρέπει να προστατευτούν αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές. Και η απειλή δεν πρέπει να είναι τέτοια εμβέλεια ώστε να αποκολέσουμε την υποστήριξη του κοινού και των πολιτών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε αυτές οι αξίες να μην λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη, στην έρευνα και στην εφαρμογή υλοποίηση των τεχνολογιών. Η ΚΑΚ υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση, αυτή τη σφαιρική ολοκληρωμένη προσέγγιση και θα συνεχίσει να είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των επιβατών. Τέταρτον, πρέπει να διεξαγάγουμε μελέτες επιπτώσεων πριν από ρυθμιστικές αλλαγές ή αλλαγές των πλαισίων, των ρυθμιστικών πλαισίων. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε αθρηστικά νέα μέτρα αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επιπλέον οι βιαστικοί, οι βιαστικοί κανονισμοί και οι βιαστικές ρυθμίσεις δεν είναι οι πιο αποτελεσματικοί ή αποτελεσματικές. Πρέπει να υπάρξει βέλτιστο πλαίσιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές και ο κοινό ε, ε, νους πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. Πρέπει να δημιουργήσουμε δυναμικό ώστε μέσω περιφερειακών πρωτοβουλειών ε, και ανάληψης δράσης να αντιμετωπιστούν οι απειλές. Να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση και γνώση των πολιτισμικών, πολιτιστικών διαφορών και θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο αυτό να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Κανένα δεν ζει απομονωμένος σε ένα νησί σε ένα στεγανό πλαίσιο χωρίς να επηρεάζεται από άλλους. Και έτσι οι ε, ενέργειες μεταφορές έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και οι ρυθμίσεις τους πάλι παγκόσμιο χαρακτήρα. Και όσον αφορά και τον, την σάρωση ε, των επιβατών αλλά και την ασφάλεια των εμπορευμάτων. Πρέπει να προαχθούν τέτοιου είδους περιφερειακές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια Στι ενέργειε μεταφορέ και την ασφάλεια των επιβατών. Το έχουμε αναφέρει και το έχουμε επαναλάβει πολλέ φορέ ο ΣΥΚΑΚ. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω ΣΥΚΑΚ. Τούτων λεχθέντων λοιπόν σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας προσφέρατε να σας προσφωνήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή τεχνική ενημέρωση αν επιτραπεί από τα χρονικά πλαίσια. Θα θέλαμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι αν περαιτέρω τεχνικές ε, αποσαφηνίσεις ε, θα ε, ζητούντο, θα προτείναμε σε μια υστερότερη φάση μια και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση μαζί σας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε ερωτήσεις σας και ελπίζουμε ότι θα χαρακτηρίσει αυτή η συνεδρίαση, θα σφραγίσει μια διαδικασία που θα συνεχιστεί στο μέλλον μαζί σας. Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, από κοινού εξ ονόματος της ΣΥΚΑΚ είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε ενδεχομένα περαιτέρω ερωτήσεις που θα είχατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την εισαγωγή και την παρουσίασή σας. Έχω αρκετούς ε, ομιλητές στον κατάλογό μου. Ελπίζω να μπορέσουμε να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας στα τρία λεπτά, ώστε να υπάρχει και χρόνος για απαντήσεις από πλευρά ΣΑΙΚΑ σε περίπτωση ερωτήσεων. Ο κύριος Δεγκράντης Πασκουάλ καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο εκπροσώπους της ε, Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας. Κατά μένα είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ. Όπως ξέρουν και οι ομιλητές μας, ε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο είχαμε μία αντίδραση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με μία έκθεση πρωτοβουλίας, στην οποία έκθεση εξετάζουμε συνολικά το όλο θέμα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. εκφράσαμε την άποψή μας για τους αρετός σώματος, ε, για τα υγρά και τα εμπορεύματα. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, έδωσε την άποψή της μέσω επιτροπολογίας, κάτι το οποίο δεν μας αρέσει και ιδιότερα. Ελπίζουμε στη συνέχεια να έχουμε και νομοθετική πρόταση, αυτό που επιθυμεί το Κοινοβούλιο, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ε, δεν μπορεί να αποξενωθούν από τις τεχνικές αποφάσεις της ε, διάσκεψης. Εγώ ως ε, συντάκτης της γνωμοδότησης έλαβα υπόψη τις μελέτες και τα στοιχεία που έχουμε ως προς τη βιωσιμότητα της διάσκεψης. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το θέμα των υγρών. Δεν θέλω να μιλάμε για περασμένα, ξεχασμένα πράγματα. Ξέρουμε ότι στις 21 Απριλίου υπήρξαν κάποιες οφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί για τα θέματα των φορολόγητων και ξέρουμε ότι διάφορα κράτη-μέλη και ερωλημένες έκαναν διαμαρτυρίες, αλλά καλό θα ήταν να σταματήσει η συζήτηση αυτή. Εμένα προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Εγώ όμως είχα κάποια ενημέρωση από τη διάσκεψη ότι υπήρχαν κατάλληλες τεχνικές ώστε να μπορέσουμε ε, να θέσουμε σε εφαρμογή εγκαίρως τους μηχανισμούς αυτούς. Θα ήθελα να μας πει η, η ΕΕΠΑ ε, εάν από τεχνολογική σκοπιάς υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως πολύ περισσότερο και νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουν να γνωρίζουν είναι κατά πόσον θα έχουμε τα κατάλληλα συστήματα για να ελέγξουμε τις ε, χειραποσκευές, ε, να δουν αν περιλαμβάνονται στερεά ή υγρά τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο ενδεχομένως και κατά πόσον οι συσκευές αυτές θα μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ ενός ε, αυλαβού υγρού και ενός υγρού που δυνητικά είναι επικίνδυνο και μπορεί να ε, προκαλέσει κάποια ε, σοβαρή ζημία επί του αεροσκάφους λάβαμε τα θετικά στοιχεία ότι η τεχνολογία προοδεύει, ότι καθημερινώς ε, οδεύουμε προς την τελειότητα για τις συσκευές αυτές, αλλά δεν ξέρω εάν ε, σήμερα μπορείτε να μας πείτε με σαφήνεια ότι το 2013 θα έχουμε τα συστήματα σε λειτουργία. Νομίζω ότι αυτό θέλουμε να γνωρίζουμε. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι το 2013 θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όσον αφορά το θέμα των σαρωτών, νομίζω ότι αντίστοιχη είναι η κατάσταση. Η ΕΒΠΑ ήδη ετοίμασε και εξέτασε κάποια συστήματα, συστήματα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ των. Θα το εξηγήσω αυτό αργότερα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ποια είναι τα κατάλληλα συστήματα και ποια όχι. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν συστήματα τα οποία θα έχουν κάποια προστιθέμενη αξία και θα μπορούν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τους κινδύνους και κατά πόσο θα έχουμε αυτά τα συστήματα ε, για να τηρηθούν και οι υποχρεώσεις μας. Τρίτη ερώτηση. Τι γίνεται με τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες όσον αφορά τις τεχνικές και τη τεχνολογία. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούμε εμείς και αυτών που χρησιμοποιούν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, και ορισμένες φορές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαρωτές σώματος γιατί απαγορεύουν αγοράζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ προσπαθήστε να τηρήσετε τα χρονοδιαγράμματα. Ο κύριος Αλκαντράουι. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εισαγωγή που παρουσιάστηκε. Τα συμπεράσματα ακούγονται πολύ καλά και θέλουμε όλοι σίγουρα να έχουμε αναβαθμισμένα επίπεδα ασφάλισης, ε, ασφάλειας, ε, διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων, ε, αναλογία σε σχέση με το κόστος και το όφελος. Όμως η πείρα στα τελευταία χρόνια τι κατέδειξε, ότι ουσιαστικά χωλένουμε και τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και τα επεισόδια. Αν κάτι συμβεί και υπάρξει κάποιο γεγονός, τότε αντιδρούμε βιαστικά και θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε ποιες επιπτώσεις έχουν οι αποφάσεις μας. Να δούμε τα κενά τα οποία δημιουργούνται, ε, πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν. Αυτό το οποίο απουσιάζει εδώ είναι μια γενική πολιτική για θέματα ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους. Δεν ξέρω αν εσείς εκπροσωπείτε και εσείς αυτή την άποψη. Θα είσαστε και εσείς υπέρ μια τέτοια ε, προσέγγισης ή μόνο θέλετε να αντιδράτε σε μηνύματα που θα αποστέλουν οι εθνικές αρχές σε εσάς όσον αφορά εντολές για κάποια δράση ή πιστεύετε ότι αμφίδρομα θα πρέπει να δράσετε, να υπάρχει δηλαδή και ενημέρωση των εθνικών αρχών από πλευρά, της, από πλευρά σας, ώστε να υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι η τεχνολογία μετεξελίσσεται και ενημερωση των εθνικων αρχων απο πλευρα της απο διαρκώς, αλλά και πριν από δύο χρόνια ακούσαμε τα ίδια και μας είπαν ότι το 2010, το 2011 λέει το αργότερο, θα είχαμε συσκευές με τις οποίες θα μπορούσαμε να ανοιχνεύουμε όλα αυτά τα ύποπτα υγρά και ουσίες και ότι έτσι οι ε, επιβάτες θα μπορούσαν ποτά παλί ή υγρά τέλο πάντων που θα χρησιμοποιούσαν για να πιούν να τα μεταφέρουν απροβλημάτιστα μαζί τους. Τώρα έχουμε μια νέα προθεσμία, 2013. Μέχρι τότε λέει θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν οι συσκευές και οι εξοπλισμοί μας. Τώρα, τούτον λεχθέντων έχω μια ερώτηση πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με την αναλογία, αναλογικότητα μεταξύ των δράσεων της ΣΥΚΑΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η αριθμιστική αρχή, υπάρχουν οι εθνικές αρχές, οι εθνικοί επαΐοντες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία απόφαση, ένα σχέδιο απόφασης. Το Κοινοβούλιο έχει ε, τώρα, θα πρέπει να έχει και δικαίωμα αρνησικυρίας όταν έχουμε 44 κράτη στην ΙΚΑΚ και έχουμε και το πλαίσιο της ε, ΙΚΑΚ, της Ρυθμιστικής Επιτροπής και το πλαίσιο των κρατών μελών, πώς όλα αυτά αλληλοσυντονίζονται. Υπάρχει ανταλλαγή που διασφαλίζεται μεταξύ των διαφορετικών απόψεων. Πώς εποπτεύεται τις συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει βέβαια ως θεματοφύλακας για τα συμβαίνουν στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενιαία εφαρμογή διατάξεων ακόμα και αν υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά εφαρμογή κάποιων πραγμάτων στα κράτη-μέλη. Τι γίνεται όμως με τα 44 κράτη-μέλη της ΙΚΑΚ. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι ή μόνο θεωρητικά υπάρχουν έλεγχοι. Thank you, Chairman, thank you. Η κυρία Φώστερ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της ΕΘΠΑ που ήρθαν σήμερα εδώ. Νομίζω ότι αυτά που μας είπαν ε, μας έδωσαν ε, τροφή για σκέψη. Καταρχάς να πω το εξής. μετά την 11η Σεπτεμβρίου παρακολουθήσαμε και εμείς πάρα πολύ ε, στην Επιτροπή μας τα όλα θέματα της ασφαλείας, το 23-20 και τα λοιπά. Ποιος είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ο στόχος μας το one-stop security. Φυσικά θα υπάρχουν κάποιοι επιβάτες που θα περνούν από την ασφάλεια ε, στη χώρα Α και μετά από τη χώρα Β εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οπουδήποτε αλλού. Και μέχρι να έχουν ολοκληρώσει το ταξίδι τους ε, θα έχουν μπουχτίσει. Ε, τα δέκα τελευταία χρόνια αυτό βλέπουμε άλλωστε να γίνεται. Άρα, ο στόχος μας τελικά ε, ποιος είναι και τι θέλει να κάνει η Κομισιόν. Υγρά πρώτα απ' όλα. Όλοι ήθελαν αυτό με τα 100 ml ε, μέχρι το 2011 να ε, πάψει να ισχύει. Πρακτικά δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Αν δει κανείς τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Αν δει κανείς τα μικρά αεροδρόμια. Καταλαβαίνω τον τύπο ΑΒΓ που λέτε, γιατί δεν έχετε και την κυκλοφορία. Δεν μπορείτε να αρχίσετε να βγάζετε, μπορείτε να αρχίσετε να κάποια αντικείμενα από τις σας και τα λοιπά. Αν δεν είναι έτοιμα οι μηχανισμοί ΔΕΛΤΑ, πώς θα εισαγάγετε αυτό το σύστημα το 2011 θα μποτιλιαριστούν τελείως οι επιβάτες. Για τρεις ώρες ε, θα περιμένουν ε, στην ουρά για να βγουν όλα τα μπουκάλια από τις αποσκευές κτλ. Ε, τέλος πάντων, το 2013 ας είναι, αλλά αφού το 2011 δεν μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά ας είναι τότε έτοιμη αυτή η μηχανισμή σε ό,τι αφορά τα είδη εξοπλισμού. Εσείς στην ιστοσελίδα σας ε, μιλάτε για τον αποδεκτό εξοπλισμό, διαφημίζετε θα έλεγα τον αποδεκτό εξοπλισμό. Είναι σαφές αυτό για τα αεροδρόμια όμως. Δηλαδή ξέρουν τι ε, εξοπλισμούς θα πρέπει, τι μηχανήματα θα πρέπει να έχουν στη θέση τους και να χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά ε, τους αρωτές σώματος, ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις εδώ και κάποιο καιρό. Και θέλω να ρωτήσω το εξή ότι ε, έχουμε τις εταιρείε που μας λένε για τους διάφορους εξοπλισμούς. Και νομίζω ότι στην Επιτροπή μας έχουμε ξεκαθαρίσει τι δεν θέλουμε παρά κάποια ιατρικά στοιχεία που δείχνουν το αντίθετο και το οποιο εχουν έχουν προσκομίσει κράτη-μέλη. Εμεί δεν θέλουμε Χ. Ούτε backscatter radiation. Κάποια κτηνοβολία διασποράς. Υπάρχουν κάποια θέματα, αυτά πρέπει να τα δούμε. Δεν θέλουμε ορισμένα πράγματα. και κάποια αεροδρόμια χαίρονται που δεν υπάρχουν αυτοί οι εξοπλισμοί έτοιμοι το 2011 γιατί κοστίζουν και πάρα πολύ. Σίγουρα για τις επιχειρήσεις βέβαια ε, ισχύει το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά όμως τους αρωτές όμως για να επανέλθω. Θέλουμε να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα. Γιατί αν ε, υπερβάλλουμε θα περνάμε όλοι από μαγνητικό τομογράφο, μήπως έχουμε καταπιεί κάτι. Και όλο και κάποτε μπορεί να συμβεί ένα συμβάν. Το θέμα είναι μέχρι που μπορούμε να πάμε. Σαρωτέ άματος ω πρόσθετο εργαλείο θα μα ικανοποιούσε, θα μπορούσαμε να το δεχθούμε. Αλλά αν είναι σωστό εξοπλισμό, δεν κοιτάς τελικά τι εξαιρέσει. Γιατί έχει νόημα να υπάρχει ένα σαρωτής σώματος όταν απαλλάσσεται ή εξαιρείται ο μισός πληθυσμός, οι έγκυες, ε, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά ή κάτι άλλο τέλο πάντων. Αν είναι σωστό ο εξοπλισμό, αν είναι εντάξει ο εξοπλισμό. ναι θα ολοκληρώσω, εάν λοιπόν είναι εντάξει ο εξοπλισμό, τότε θα πρέπει λογικά να μπορεί να περάσει οποιοδήποτε από αυτό το σαρωτή, ανεξαρτήτως ηλικία, ιατρικής ε, κατάστασης, εάν είναι σωστός εξοπλισμός. Μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε ε, ένα πρόσθετο εργαλείο ή το σαρωτή σώματος που θα είναι χρήσιμος. Αν είναι θελοντικό και αν κάποιος μπορεί να εξαιρεθεί, έχει νόημα τελικά. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις μου και ένα τελευταίο σχόλιο. Με την Άσα τι σχέσεις έχετε, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΦΠΑ για την ε, παρουσίαση και να κάνω μια παρατήρηση. Βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι το θέμα της ασφάλειας και ο καθορισμός αντικειμενικών κανόνων, γιατί η αντίληψη της ασφάλειας είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα, το βαθμό της απειλής, τη γεωπολιτική θέση ενώ στην προστασία ε, είναι λίγο πιο αντικειμενικά τα στοιχεία. Ε, αν θέλετε μου απαντάτε ε, πόσο περίπου εκτιμάτε ότι είναι το αποδεκτό επίπεδο κάποιου σφαλμάτων για τα υγρά τύπου CD. Και όταν έχει υπάρξει σφάλμα δηλαδή false alarm κατά κάποιο τρόπο, τελικά τι γίνεται. Ξαναπερνάει από έλεγχο και μετά κενώνεται η περιοχή και φέρνουν στους πυροτεχνουργούς. Τι γίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία γιατί ε, αν έχουμε συνέχεια false alarm και μετά ξεκινάνε ολόκληρες διαδικασίες ε, που παίρνουν ώρα, ξέρουμε ότι θα μπλοκαριστεί η κίνηση στο αεροδρόμιο. Και σε ό,τι αφορά ε, τις δυνατότητες ανείχνευσης, Έχουμε το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, μια αρχή που μπορεί να χρησιμοποιούν ε, οι ορισμένοι σαρωτές. Υπάρχουν τα διάφορα συστήματα, το backscatter που δεν θα θέλαμε και αυτό ε, με τα που θα θέλαμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν του σαρωτές ασφαλείας, έχουμε κάποια ιδέα, θα γίνουν δοκιμές και πότε. Thank you, Mrs. three minutes, please. Κυρία Γιάλα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους υπευθύνου τη ΕΔΠΑ για την παρουσίασή τους και θα ήθελα να κάνω και τρεις μικρές παρατηρήσεις. Καταρχάς μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα ποιοι συμμετέχουν ε, στον καθορισμό των προτύπων. Εντάξει, εμπειρογνώμονε, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν ερωτήσει και προ του τελικέ χρήστε και τους επιβάτες, ε, διότι το πρώτο σας σύνθημα ήταν να έχουμε ε, κανονική, πραγματική ασφάλεια ε, βάσει και των απαιτήσεων των επιβατών. Τι κάνετε γι' αυτό. Επίσης, πώς περνάμε από τη θεωρία των δοκιμών που κάνετε εσείς στην πραγματικότητα των αεροδρομίων με επιβάτες, ε, μικρά αεροδρόμια που λειτουργούν εποχιακά ε, και τι γίνεται με τις προθεσμίες. Εσείς μας λέτε ότι η κατηγορία D που είναι αυτή που θα μας επιτρέπει να μην ανοίγουμε τις χειραποσκευές και να κάνουμε τον έλεγχο και είναι αυτό που δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα στα, στους επιβάτες ε, είναι αυτή που θα δοκιμάσετε από το 2011 και τούδε. Από τη στιγμή που θα γίνουν οι δοκιμές μέχρι να ολοκληρωθούν και να εγκριθούν, τι προθεσμίες προβλέπονται, εάν φυσικά τις γνωρίζετε. Και τέλος, ε, Αναφερθήκατε στην ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα για τους επιβάτες. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, όχι μόνο για το ποιους ταξιδεύουν υπερατλαντικά ή όχι, αλλά και στα ίδια τα κράτη-μέλη δεν αναφέρομαι μόνο στα υγρά εκρηκτικά, αλλά στους αρωτέ εν Υπάρχουν αεροδρόμια στα οποία πρέπει να βγάλει άλλο τον υπολογιστή του ή ε, κάποιοι τον υποχρεώνουν να τον ανοίξουν κιόλα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν, πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις διαφορές που κάθε φορά συγχαίουν όλο και περισσότερο τους ε, ε επιβάτες, ε, νιώθουν ότι ε, τους αντιμετωπίζουν ε, ε, επιθετικά. Πώς μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε με τους επιβάσεις, επιβάτες και τι συγκεκριμένες ε, συστάσεις μπορείτε να κάνετε, διότι υπάρχει πλήρη σύγχυση και εκνευρισμός ε, και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που δημιουργεί όλο και μεγαλύτερο χάος και μεγαλύτερη αίσθηση ανασφάλειας. Κύριος δεν θα αφαιρέσετε το χρόνο από το χρόνο παρέμβασή μου, έτσι. Και από μένα ευχαριστώ θερμά πρέπει να πω για την εισήγησή σας και για την προσφορά σας ενδεχόμενα αυτή τη συνεδρία και κλεισμένων των θυρών να την συνεχίσουμε. Παρότι είμαστε πολιτικοί, θα παραμείνουμε πολιτικοί και δεν θα γίνουμε πραγματογνώμονες παρόλα αυτά. Είπατε κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να χαιρετήσω. Αξιολόγηση επιπτώσεων πριν από την υλοποίηση. κοινό νου που πρέπει να πριτανεύσει, διεθνείς συγκυρίες που πρέπει να αναγνωρίσουμε και προσδοκίες των επιβατών. Αν αυτά τα είχαμε πάντα παντού, τότε διαφορετικά θα συζητούσαμε τα πράγματα σήμερα. Τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω. Πρώτον, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αν το αβγ ή δ μέσα στο σύνολο των διαφορετικών σαρωτών σώματος λειτουργούν ή δεν λειτουργούν, διότι δεν έχουμε το α και το Β, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει το Γ και το Δ. Και δεν θέλουμε κανένα αεροδρόμιο να προκληθεί να δαπανίσει περιτά κονδύλια ώστε μετά από ένα-δύο χρόνια να αποκτήσει εξοπλισμό που θα είναι χρήσιμος και για τους επιβάτες επιτέλους. Θα μπορούν να αφήνουν στη χειραποσκευή τους τα υγρά τους και έτσι να σαρώνονται και να περνούν από τον έλεγχο. Και γι' αυτό η ερώτησή μου, όταν ακούω ότι το ΔΕΛΤΑ θα ξεκινήσει τέλη 2011, δηλαδή 17 μήνες πριν από τα τέλη Απριλίου 2013, βλέπετε μια ρεαλιστική πιθανότητα, ευκαιρία οι σαρωτές ΔΕΛΤΑ ...στην ημερομηνία εκείνη να μπορέσουν να εισαχθούν ή όχι. Δεύτερο ερώτημα. Και μετά επαρκούμε σε αυτά για τους σαρωτές σώματος. Διάβασα ότι τώρα μετά την απόφαση θα έχουμε εφαρμογή, υλοποίηση type testing programs τυποποιημένων προγραμμάτων ελέγχου και είπατε ότι οι πληροφορίες που στα εθνικά, στα κράτη-μέλη που είναι διαθέσιμα από στην Ολλανδία για παράδειγμα θα χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τα αποτελέσματα που έχετε σε σχέση με τη Γερμανία. Εγώ είμαι από το Αμβούργο. Οι σαρωτές σώματος όταν πάνω από 100 επιβάτες ε, ε, είναι παρόντες για, ένα, για μια πτήση δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διότι δεν επαρκεί ο χρόνος. Είναι διαφορετικές συσκευές αυτές. Τι θα γίνει με αυτές. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια για την αποτελεσματικότητα και να υποβάλλετε κάποια σύσταση για συγκεκριμένους τύπους αυτών των συσκευών. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε πολύ σύντομα. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι η έλεγχη επιβατών από 98,5% θέλουμε να βελτιωθούν σε 99%. Στην έκθεση του συναδέλφου Πασκουάντε Γκράντες έχει ε, διατυπωθεί ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μια συγκεκριμένη προβληματική που αντιμετωπίζουμε. Είναι οι συνδυασμένες μεταφορές επιβατών και αγαθών και εμπορευμάτων. Και στον τομέα των εμπορευμάτων ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια, σίγουρα. Και αυτό όχι μόνο οι δοκιμασίες το καταδεικνύουν που πριν από τόσους μήνες, ας το πω έτσι, έγιναν, αλλά η αρχή της ε, ασφαλούς αποστολής και της πιστοποιημένης ασφαλούς αποστολής που ισχύει εξακολουθεί να είναι προβληματική η κατάσταση. Εκεί έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα λέγοντας ότι πρέπει τα εμπορεύματα, τα αγαθά να εξετάζονται ιδιαίτερα, να ελέγχονται ιδιαίτερα όχι μόνο με ακτίνες χ αλλά για την ανείχνευση εκρηκτικών με οποιασδήποτε μεθόδους υπάρχουν. Το έχετε δει αυτό. Το θεωρώ θεμελιώδου σημασία σημείο για την ασφάλεια συνολικά των εναερίων μεταφορών που θέλουμε να βελτιωθεί η ασφάλεια αυτή. Thank you. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ε, και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η παρουσίαση που κάνετε και η συζήτηση που ακολούθησε. Κάποιοι ε, συνάδελφοι ανέφεραν κάποια θέματα, κάτι το οποίο εμένα έτσι ε, μου κάνει εντύπωση είναι, δεν ξέρω κατά πόσον ε, η ΕΔΠΑ ε, έχει θέσει κάποια συγκεκριμένα πρότυπα για τους σαρωτές. Αν υπάρχει ένα είδος βίβλου δηλαδή, κάποια πρότυπα, κάποιες προδιαγραφές για τους σαρωτές. Θα με ενδιαφέρε να μου απαντήσετε. Επίσης στην παρουσίασή σας είπατε ότι συνήθως αν κάποιος νομοθετήσει γρήγορα θα νομοθετήσει άσχημα. Δεν διαφωνώ, αλλά αν κάποιος, πει ε, κάποιος θα πρέπει να το πει στα κρατη αυτό. Γιατί πολλές φορές τα κράτη-μέλη ευθύνονται για γρήγορη άρα και κακή ενδεχομένως νομοθεσία. Αν κάτι γίνει αμέσως ε, σπέβδω να κάνουν κάτι και τελικά επανεφεύρουμε τον τροχό, επανεφευρίσκουμε συνέχεια τον τροχό και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν η ΕΔΠΑ ε, ουσιαστικά ασκεί κάποιε πιέσει στα κράτη-μέλη για να μην ε, σπέβδουν ε, με υπερβολική βιασύνη. όλα αυτά τα οποία οδήγησε σε όλη αυτή τη φασαρία τον Απρίλιο είναι ότι τελικά οι Ηνωμένε Πολιτείε στην τελευταία στιγμή ε, ανέκτουσαν πρίμα και δημιούργησαν, άλλαξαν άποψη και δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει κανείς που μιλάει με τις ΕΠΑ, υπάρχει συνεργασία. Και δεν εννοούμε ότι αν, πείτε, αν πούνε στη ΣΥΠΑ πηδήξτε, εμεί θέλουμε να δούμε απλά πόσο ψηλά πρέπει να πηδήξουμε εδώ στην Ευρώπη. Όχι, λέω, υπάρχει συνεργασία, πραγματική συνεργασία για να μην επαναληφθεί και η κατάσταση του φετινού Απριλίου. Το τελευταίο σημείο είναι το εξή. Φαίνεται ότι στην Επιτροπή μας, το καταλάβατε αυτό, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την προθεσμία του 2013, ότι θα τηρηθεί η προθεσμία. Αυτή την ε, δυσπιστία νομίζω δεν μπορείτε να μας την καταλογίσετε. Εμείς θέλουμε από τεχνικής πλευράς να ξέρουμε αν είναι εφικτό ναι ή όχι. Γιατί αν είναι, άντε ας το τελειώνουμε το θέμα. Πάνω σε αυτό νομίζω χρειαζόμαστε απαντήσεις από εσάς. Και το εντελώς τελευταίο θέμα, δοκιμές. Θέλω να σας πω ότι ναι, καταλαβαίνω την ανάγκη για εργαστηριακές δοκιμές. Αλλά στα αεροδρόμια είναι εκεί που πρέπει ουσιαστικά να γίνουν οι δοκιμές. Πόσο λοιπόν ποσοστό είναι οι δοκιμές σας στα αεροδρόμια σε σχέση με τις εργαστηριακές δοκιμές. Ο κύριος Μπόλτιν από την Κομισιόν ε, αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να λάβει το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο αλλά για κανένα δύο λεπτά για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Θα είμαι αυστηρός με την Επιτροπή όσο υπήρξα και με τα μέλη της Επιτροπής, ορισμένα από αυτά. Sorry. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποκλίνομαι στην αυστηρότητά σας. Καταρχάς, ε, χαιρετίζω τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι πολύ σχηδής ε, και είναι και πολύ χρήσιμη η συνεργασία αυτή. Όσον αφορά τα καθορισμένα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρότυπα για δοκιμές και επιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και τους διαβουλευόμαστε για όλα τα σημεία αυτά. Είναι πολύ ε, καλή αυτή η συνεργασία, αλλά η δουλειά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειροσωμοσύνη. Δεν θέλουμε να αλληλοεπικαλύψουμε ε, τις εργασίες της ε, Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ίσα ίσα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, γνώσεις τους. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εφαρμόσουμε την επιθυμία της Επιτροπής να επιτύχουμε το στόχο για την ασφάλεια. Έχουμε μία συνεδρίαση το Σεπτέμβριο, ώστε όλες οι πλευρές να προσπαθήσουμε να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο για τις δοκιμές. Οι κατάλληλες δοκιμές συνεχώς είναι ο κατάλληλος τρόπος για να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη φορά. Παρεπιπτόντως ε, θα γίνει και μια αναθεώρηση στα μέσα του 2012 για να δούμε κατά πόσον η τεχνολογία αρχίζει να λαμβάνει την κατάλληλη μορφή για να αποφύγουμε την ίδια παταγώδη αποτυχία που είχαμε φέτος. Τα όσα είπε ο κύριος Ελκαντράουι και τον τρόπο που εμείς αντιδρούμε. Ε, αυτό ειλικρινώς είναι ε, κομμάτι του παιχνιδιού. Ε, αντιδρούμε στις δράσεις κακών ανθρώπων και εξορισμού αντιδρούμε απλώς και μόνον. Προσπαθούμε όμως να έχουμε και πρόληψη και να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη τεχνολογία και τα κατάλληλα μέσα για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών μας. Όσον αφορά τη χρήση των νέων μοντέλων ασφαλείας, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην ε, Σιγκαπούρη με την ΕΔΠΑ και έχουμε το ίδιο όραμα με την ΕΔΠΑ. Θέλουμε να προχωρήσει το ζήτημα αυτό και θέλουμε να το συζητήσουμε με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην έκανα κατάχρηση του χρόνου που μου δώσατε. Τρία δευτερόλεπτα λιγότερο μιλήσατε κύριε Μπόλτον. Καλός ο χρόνος σας από την ΕΤΠΑ. Δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Αν θέλετε να απαντήσετε λοιπόν σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν, έχετε το λόγο. Έχουμε 10 λεπτά λοιπόν ε, περίπου για να ξέρετε πόσο χρόνο έχετε να μιλήσετε. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε 10 λεπτά, αλλά τόσο χρόνο διαθέτουμε δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ετέθησαν πολλά ερωτήματα από διάφορε οπτικέ γωνίες. Θα απαντήσω καταρχάς στα ερωτήματα του κύριου Τεγκράντες, αλλά και στο δικό σας κύριε Πρόεδρε, που ήταν πιο γενικού χαρακτήρα. Και στη συνέχεια θα συμπληρώσουμε εγώ και ο συνάδελφος ε, με στοιχεία απάντηση ε, για τις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που μας ε, θέσατε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Επιτροπή σας και ιδιαίτερα τον κύριο Τεγκράντες για την έκθεση για τους αρωτές σώματος που μας βοήθησε τα μάλα. Βέβαια πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για τους αρρώντες αλλά έχουμε μια σημαντική βάση εργασίας για ένα θέμα που δεν είναι μόνο τεχνικό, έχει και πολιτική ε, υφή για τα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και τώρα έχουμε μια σαφή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τα υγρά, Το πρώτο ερώτημα ουσιαστικά ήταν αν υπάρχουν σήμερα κατάλληλα συστήματα από τεχνολογικής πλευράς και ποιες πιθανότητες υπάρχουν να τηρηθεί η προθεσμία του 2013. Λοιπόν, θα τα πω ξεκάθαρα. Άκουσα κάποιον βουλευτή, συνάδελφό σας, τον κύριο Φλέκενστάιν συγκεκριμένα, που μιλάει για τους εξοπλισμούς τύπου Α και Β, που λέει ότι δεν επιτρέπουν να γίνουν πολλά πράγματα και συμφωνώ απόλυτα. Ο τύπος Α ελέγχει υγρά με δειγματοληψία. Φανταστείτε να έχουμε ένα μπουκάλι ουίσκι πεπαλαιωμένου ή μπορντό και να πρέπει να κάνουμε δειγματοληψία. Πάει το προϊόν, καταστράφηκε. Άρα δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ο τύπος Β είναι καλύτερος, αλλά πρέπει να δούμε αν αυτό διευκολύνει Ουσιαστικά κάθε φιάλι, κάθε φιαλίδιο το ελέγχουμε ένα προς ένα. Ουσιαστικά δηλαδή γίνεται ό,τι γίνεται μέχρι, μέχρι σήμερα που βγάζει ο επιβάτης ε, τα υγρά τα οποία δεν μπορούν να δοκιμαστούν. Αύριο μπορούν με να δοκιμαστούν αλλά και γι' αυτό θα χρειάζεται χρόνος. Και αν έχουμε και τον, ε, το υψηλό επίπεδο των ε, λάθο συναγερμών καταλαβαίνετε ότι καθυστερούμε πολύ τις διαδικασίε. Γι' αυτό πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεώρησαν ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα τους επέτρεπε να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με το σημερινό για τη σήμερα το επίπεδο ασφάλειας για τα υγρά είναι εγγυημένο λόγω του μικρού όγκου που επιτρέπεται. Οι εκρηκτικές ύλες είναι αποτελεσματικές ανάλογα με το μέγεθος ε, τη, μάζα ή τον όγκο τους. Επομένως, περιορίζοντας τη μάζα και τον όγκο, περιορίζουμε τον κίνδυνο. Αν αύριο απελευθερώσουμε τον όγκο, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε μόνο ε, μια μικρή ποσότητα φιαλιδίων, ε, μπουτικαλιών κτλ. Καταλαβαίνετε το επίπεδο ασφάλειας δεν θα είναι το ίδιο. Και γι' αυτό σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου σίγουρα ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνο σε σχέση με κάποια χρόνια πριν. Και εγώ, οι Γάλλοι γενικά, που έχουμε ε, βρισκόμαστε σε πόλεμη σύρρηξη με τη Λιβύη, παραδείγματο χάρη που κατέστρεψε ένα αεροπλάνο μα πριν από κάποια χρόνια, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και βέβαια και η κοινή γνώμη έχει σημαδευτεί από όλα αυτά. Ε, και την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όλα αυτά τα ζητήματα. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και σε πολλέ άλλε χώρε. Και αυτό εξηγεί το ότι θεωρήσαμε ότι είναι άσκοπο ε, να κατεβάσουμε τώρα ε, τον πύχη και να μην είμαστε τόσο προσεκτικοί. Έχουμε λοιπόν τον τύπο Δέλτα και εκεί έχουμε εστιάσει. Γιατί πρώτα απ' όλα γιατί θα σημάνει μια πραγματική πρόοδο σε σχέση με τον επιβάτη που δεν θα χρειάζεται πλέον να βγάζει όλα τα υγρά που μεταφέρει μαζί του. Θα περνά ε, τη χειραποσκευή του όπως σήμερα από τον νήματα και έπειτα όταν θα βγαίνει ε, από τη, τον Νιμάντα θα ελέγχεται χωρίς να πρέπει να τον αδειάσει το μισό, ε, τη μισή βαλίτσα. Θα είναι πιο γρήγορη διαδικασία λοιπόν. Άρα με το ίδιο επίπεδο με την ίδια ουράν θέλετε, τον διορθμό επιβατών περιμένει στην ώρα, θα ελέγχουμε πολύ περισσότερο τις αποσκευέ. άρα θα βελτιώσουμε το επίπεδο ασφάλεια, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ευκολία μετακίνηση των επιβατών. Επίσης, ο ίδιος είναι ο στόχος στην ΕΔΠΑ με αυτόν τις Κομισιόν και της δικής σας Επιτροπής, δηλαδή να λειτουργούν καλά τα καταστήματα αφορολογή των ειδών, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ρουλιμενικής οικονομίας, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με σεβασμό σε αυτή την αρχή της ασφάλειας. Τώρα, επόμενο ερώτημα, θα είμαστε σε θέση να τηρήσουμε την προθεσμία του 2013. Αν με επιτρέπετε, δεν θα πρέπει να μας κάνετε να παίξουμε ένα ρόλο που δεν έχουμε. Δεν είμαστε αυτοί που θεσπίζουμε τα χρονοδιαγράμματα, ούτε εμείς κατασκευάζουμε κάποιο μηχάνημα. Όσο εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πιέσουμε τους ε, βιομηχάνους, ε, τους κατασκευαστές να ετοιμάσουν τα μηχανήματα το συντομότερο δυνατό. Εμείς είμαστε σε θέση να μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να κάνουμε τις δοκιμές και τις εργαστηριακές και μετά ε, τις επιτόπιες δοκιμές σε, στα αεροδρόμια. Αλλά εργαζόμαστε με τους εξοπλισμούς που ε, μας διαθέτουν. Και όπως είπε ο κύριος Ρικέ, έχουμε υπόψη μας και τη σημερινή απειλή, αυτό το πλαίσιο. Αλλά αυτό ε, μεταβάλλεται. Είναι ρευστή η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πολλά ήταν τα ερωτήματα για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτα απ' όλα παρακολουθούμε, είναι συνεχείς οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε χρόνο έχουμε συνάντηση, μάλλον δύο φορές το χρόνο συναντόμαστε με τους ε, ομολόγους μας από τις ε, ΗΠΑ, μία φορά στην Ευρώπη, μία φορά στην ε, ΣΥΠΑ. Και με το TSA και με το ε, DGA. Δηλαδή βλέπουμε όλους τους ε, φορείς για την ασφάλεια της αεροπορίας και εναέρειες επιχειρήσεις, ε, ασφάλεια ε, αεροπλοείας κατά πολέμηση τρομοκρατίας και περιβάλλον. Αυτές είναι οι τρεις ε, συνιστώσεις στις οποίες έχουμε συνεργασία, διαρκή και σταθερή. Προσπαθούμε να συντονιστούμε, αλλά κάθε ομάδα είναι ξεχωριστή. Κυρίαρχη θα έλεγα. Και ο πρόεδρος μας έχει πει πολύ ξεκάθαρα ότι οι κυβερνήσεις αντιδρούν ε, σε συνάρτηση με τα γεγονότα. Μπορούμε να καταλογίσουμε στις κυβερνήσεις. Ότι κάποιες φορές αντιδρούν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά τι θα λέγαμε αν δεν είχαμε προσπαθήσει να ε, διδαχθούμε από μία απόπειρα. Και αν μετά ε, βλέπαμε μια επόμενη απόπειρα να έρχεται χωρίς να έχουμε αντλήσει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις που η κυβέρνηση καλείται να προβεί σε αποφάσεις ε, όταν όλα είναι ασαφή και αβέβαια. Γνωρίζουμε ότι δημιουργούμε προβλήματα σε άτομα απόλυτα αθώα, που, ακίνδυνα, που δεν φταίνει σε τίποτα, αλλά καταλαβαίνετε τι καταστροφικές επιπτώσεις θα είχαμε αν δεν, κάναμε, ε, αν δεν παίρναμε αυτά τα μέτρα. Σίγουρα δεν είμαστε στην τελειότητα σήμερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια συνέπεια, ε, συνεκτικότητα των μέτρων ε, που έχουν θετήσει τα κράτη που συμμετέχουν στη GAC. Και νομίζω ότι υπάρχουν κοινέ θέσει μεταξύ των κρατών μελών. Ένα άλλο ερώτημα είχε να κάνει με την λειτουργία της ΕΔΠΑ. Έχουμε ουσιαστικά 44 κρατημέλη, όλα τα κρατημέλη της Ένωσης, αλλά περισσότερα από αυτά. Άρα είμαστε ευρύτεροι ε, στη σύνθεσή μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδηγίες που θεσπίζουμε είναι οδηγίες που τις δέχονται ελεύθερα τα κράτη-μέλη μας. Δεν έχουμε ρυθμιστικές εξουσίες και είναι προφανές ότι για τα κράτη-μέλη της Ένωσης που είναι και μέλη της ΕΔΠΑ οι κανόνες που πρέπει να τηρούν είναι οι κοινοτικοί κανόνες. Πάντως όσο ευρύτεροι είναι οι κανόνες, τόσο πιο αποτελεσματικά θα είναι τα μέτρα, γιατί τα αεροπλάνα πετούν μακριά, άρα η, καλύτερη, μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη είναι ό,τι καλύτερο. Άρα καλό θα ήταν διεθνώς να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε σε επίπεδο των 44 δηλαδή κρατών, να προωθήσουμε κανόνες που κάποιοι είχαν σχεδιαστεί σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά πρέπει να διδαχθούμε και από τις εμπειρίες άλλων χωρών μεταξύ των 44. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν νομοθετική ρυθμιστική εξουσία. Δεν είμαστε τέ, φορέας τέτοιο, δεν είμαστε σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Αυτό είναι προφανές. Σε ό,τι αφορά τους αρωτές σώματος τώρα. Το μήνυμα το λάβαμε, το λάβαμε ξεκάθαρα ότι την ότι την κτηνοβολία πρέπει να την αποφύγουμε. Αυτή την επιλογή την είχαν κάνει και κάποια κράτη που είχαν επιλέξει το μιλιμετρικό σύστημα το οποίο δεν έχει κίνδυνο ακτινοβολία. Είπα, έκαναν μια διαφορετική επιλογή. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν και του δύο ε, τύπου και τα δύο συστήματα. Και την ακτινοβολία οπισθοσκέδαση ε, και τη, το μιλιμετρική τεχνολογία. Οι αναλύσει ε, που δείξαμε δείχνουν ότι η οπισθοσκέδαση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο. Βέβαια, είναι λογικό να ακολουθήσουμε και δεν θα έχουμε κανένα διστάγμα να το κάνουμε τις δικές σας ε, συστάσεις σε ό,τι αφορά τους ε, σαρωτές σώματος εντύσσεως της ακτινοβολίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την, ε, τον, τον έλεγχο ε, που γίνεται με τα χέρια, αν ε, η ψηλάφιση γίνεται επαρκώς μπορεί να αποφέρει πολύ καλά αποτελέσματα, αν δεν γίνεται καλά δημιουργεί προβλήματα. με το αυτόματο, με το αυτόματο λιγότερο του σαρωτών σώματος θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, ελπίζοντας βέβαια να έχουμε και έναν τρόπο αποφυγής ε, της ε, καταπάτησης της ιδιωτικής σφαίρας. Ε. Δυστυχώ διακόπτει ο πρόεδρο. Ολοκληρώνεται. Ναι, ολοκληρώνεται. Ήταν το τελευταίο σημείο. Έλεγα ότι ο αυτόμα, η αυτόματη λειτουργία, αν τον βάλουμε στο automatic mode, το σαρωτή δεν θα είναι σίγουρα τόσο αποτελεσματικό. Γιατί τέλο πάντων πολλά εξαρτώνται και από τον ανιχνευτή και από το σύστημα που αναλύει την εικόνα αλλά φαντάζομαι ότι θα προοδεύσει τεχνολογία. Ε, αυτά είχα να σας πω, έτσι λίγο ανακατεμένα. Δεν ε, τήρησα τη σειρά των ερωτημάτων, αλλά νομίζω ότι με το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου καλά τα πήγα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φώστερ κάτι θέλει επί της διαδικασίας. Θα πρέπει να είσαι πολύ σύντομη, Τζάκη, γιατί έχουμε και τον Ούγκρο Υπουργό εδώ. Ένα σημείο θέλω να θίξω, γιατί έγιναν πολύ έντονε συζητήσει για την ακτινοβολία σα και εσεί έχετε την άποψή σα, αλλά έχουμε και εμεί την άποψή μα και δεν συμφωνούμε εν γέννη με αυτά που λένε ε, οι άνθρωποι τη ιατρική επιστήμη που λένε ότι δεν υπάρχει καμία επιρροή για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η όλη διαδικασία εάν εισαχθεί ένα σαρωτή σώματο και είναι τέτοια τεχνολογία ώστε να, υπάρχει, να μην υπάρχει κανένα ερωτηματικό για θέματα υγεία και να μην εξαιρείται κανεί από αυτά, τότε σαφώ είναι η σωστή κατεύθυνση αυτή. Ιδάλω, ε, ο μισό πληθυσμό θα εξαιρείται και οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα παίρνουν από του σαρωτέ. Αυτό είναι το θέμα που θίξιμα και αυτό είναι το θέμα της ε, ακτινοβολίας ε, οπισθοσχέδεση, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Αυτό που θέλουμε είναι ένα σύστημα ενιαίο για όλη την Ευρώπη ώστε να υπάρχει συνέπεια και συνέπεια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, μπορεί στο ένα αεροδρόμιο να υποχρεώσει να βγάλει τα παπούτσια σου και στο άλλο αεροδρόμιο να μην υποχρεώσει να βγάλει τίποτα και όλα να είναι στο ίδιο κράτο μέλο. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι και θέμα συνέπεια. Ευχαριστούμε λοιπόν ε, του ε, κυρίου από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτική Αεροπορία που ήρθαν εδώ σήμερα και μα έκαναν αυτή την παρουσίαση και θα δεχτούμε την προσφορά σα να υπάρχει ένα συνεχή διάλογο μεταξύ Ευρω... Επιτροπής ε, ε, Μεταφορών και Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας. Νομίζω ότι θα αφοληθούμε και οι δύο από αυτή την ανταλλαγή απόψεων και εκτιμούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ότι θα πρέπει, ε, στις οποίες θα πρέπει να κάνουμε συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών, διότι υπάρχουν και θέματα εμπιστευτικότητας και ασφαλείας. Δεν θα είναι πρόβλημα αυτό για μας, μπορούμε να το διοργανώσουμε. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία και την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να περάσουμε τώρα απευθείας στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βόλνερ, τον Υπουργό Μεταφορών της Ουγγαρίας και προεδρεύοντα το τελευταίο εξάμεινο στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Ζητώ συγγνώμη που σας ε, άφησα να περιμένετε. Έχετε το λόγο. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας για να κάνουμε τη συζήτησή μας. Ε, αν μπορείτε λοιπόν να κάνετε μια παρέμβαση περίπου 15 λεπτών ε, προκαταρκτικά και από εκεί και πέρα να δώσουμε το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι μια θεμελιώδους σημασία συγκυρία για την Ουγγαρία. Όταν ανέλαβε η Ουγγαρία την ανακυκλούμενη Προεδρία του Συμβουλίου για πρώτη φορά σε αυτή μας τη θητεία. Προσβλέπαμε και αναμέναμε αυτό το έργο με μεγάλες προσδοκίες και συμμετείχαμε στην προπαρασκευή του προγράμματος για τις μεταφορές και σε σχέση και με την τις προηγούμενες σε σχέση με την πολιτική για τις μεταφορές, στο πρόγραμμα της Προεδρίας μας, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για μια ανταγωνιστική και ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση για την αηφορία, ένα αηφόρο σύστημα μεταφορών για την Ευρώπη προσπαθώντας να επιτύχουμε τους στόχους της Προεδρίας μας μέσα στο πλαίσιο μιας φιλο ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πολιτικής, φιλικής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πολιτικής. Θέσαμε φιλόδοξους στόχους ε, όσον αφορά την πολιτική για τις μεταφορές ως Προεδρίας και με επιτυχία καταφέραμε να επιτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε τους περισσότερους στόχους μας. Είμαι πισμένος ότι δεν θα είχαμε καταφέρει να πετύχουμε χωρίς την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, ιδιαίτερα χωρίς την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βέβαια. Για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον επικοδομητικό τρόπο στη συνεργασία και για την υποστήριξη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις προς τις προτάσεις της Ουγγρικής Προεδρίας. Οι κοινέ μας προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να προσδώσουν επαρκείς αποτελεσματικές απαντήσεις στα θέματα των μεταφορών για την Ευρώπη, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας, τονώνοντας τα θέματα μεταφορών και προωθώντας την ευημερία, υποστηρίζοντας την περαιτέρω διεύρυνση της ευημερία των πολιτών μας. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας δώσω σύντομα μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων εν περιλήψη της Ουγγρικής Προεδρίας όσον αφορά την πολιτική για τις μεταφορές το πρόγραμμα της Προεδρίας τα χαρτοφυλάκια αυτά τα ενέταξε σε δύο κυριότερους στόχους, αηφορία και ολοκλήρωση αφενός και αφετέρου ασφάλεια και αηφορία, κυρίως ασφάλεια. Όσον αφορά την ασφάλεια και τα παντελή θέματα ασφάλειας και ολοκλήρωσης, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στο χαρτοφυλάκιο για την αναθεώρηση και αξιολόγηση των τεκτενομένων όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου στο Γκέντελε της Ουγγαρίας ήταν ένα από τα κύρια κλειδιά στις εκδηλώσεις της Ουγγρικής Προεδρίας. Σε αυτή την συνεδρίαση, σε αυτή τη σύνοδο επικεντρωθήκαμε στο μέλλον των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ιδιαίτερα στα θέματα σχεδιασμού των δικτύων και στα θέματα χρηματοδότησης των δικτύων. Τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου στο Γκέντελε οι προσδοκίες των κρατών μελών που έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτές όσον αφορά και το σχέδιο νομοθετικής δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάχθηκαν στα συμπεράσματα του, της Προεδρίας από κοινού και με την τελευταία ανακοίνωση που δώσαμε προς τον τύπο ως Προεδρία. Σαν αποτέλεσμα αυτής της άτυπης συνάντησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε διμερείς διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη για το γενικό πλαίσιο αλλά και τον πυρήνα αυτών των σχεδίων. Αυτές οι διαβουλεύσεις από κοινού με τα συμπεράσματα συστάσεις της Προεδρίας οδήγησαν στην, ε, σε ένα πλαίσιο νομοθετικό και προτάσεων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών το Σεπτέμβριο. Επίσης ε, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική όσον αφορά το λευκό βιβλίο ήταν ένα άλλο στοιχείο στρατηγικής σημασίας σημαντικό για την Ουγγρική Προεδρία. Προχωρήσαμε και συμμετείχαμε σε συζητήσεις ουσιώδους χαρακτήρα με το Συμβούλιο και όσον αφορά και την προπαρασκευή λήψης αποφάσεων καθώς επίσης λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τη δημοσίευση του Λευκού Βιβλίου. Είχαμε μια ουσιώδη συζήτηση επ' αυτών και οδηγηθήκαμε και στην περίληψη το, στα συμπεράσματα από πλευράς της Προεδρίας. Τα κράτη-μέλη χαιρέτησαν καλοδέχτηκαν τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρότι δεν ενέκριναν όλα τα επιμέρους στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών έτσι όπως είχαν πρώτα παραταθεί θέματα προτεραιότητας. Τα κράτη-μέλη τόνισαν τα θέματα έρευνας και καινοτομίας στην πολιτική για τις μεταφορές, την αποτελεσματική διασύνδεση και αλληλεξάρτηση των θεμάτων ε, επιμέρους ε, ε, συνιστοσών και παραμέτρων, την ολοκλήρωση ενός ενιαίου πλαισίου μεταφορών την ανάπτυξη των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και της δυνατότητας συγχρηματοδότησης ώστε να διασφαλιστούν οι υποδομές στις ε, μεταφορές καθώς επίσης και ένα εθνικό τοπικό περιφερειακό πρόγραμμα δράσης ε, για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, καθώς επίσης και οδικές, οδικό χάρτη για τις προτάσεις όσον αφορά την FEE, τα e συστήματα ε, για τις μεταφορές και από κοινού με τις περιφερειακές προτάσεις ε, των κρατών μελών αυτή η περίληψη αυτή η επισκόπηση δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια επαρκή, επαρκώς πλήρη εικόνα για το ποιες είναι οι θέσεις των κρατών μελών και για το πώς διατυπώνονται, σε ποιο πλαίσιο διατυπώνονται οι προτάσεις. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία, με βάση την πολιτική συμφωνία που επετέχθη με την ε, ε, ειδική πλειοψηφία υπό την Βελγική Προεδρία διαπραγματευτήκαμε, κάναμε τις ε, αναγκαίες διαβουλεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την δεύτερη ανάγνωση αυτών των θεμάτων πέτυχε τους στόχους της η Προεδρία. Διαπραγμάτευση επί των θεμάτων που ε, λίμναζαν από το 2008 επετέφθη, ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις και επετέφθη σε δεύτερη ανάγνωση συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την αναθεώρηση της οδηγίας στη συνεδρίασή του της 7ης Ιουνίου 2011 και αυτή η νομοθεσία είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της χρησιμοποίησης της εφαρμογής της αρχής ο πληρώνει όσον αφορά τα συναφή θέματα που άπτονται των μεταφορών. Και θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Αλκαντράουι που ήταν ο εισηγητής για αυτό το χαρτοφυλάκιο από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε όπως επίσης και τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών τον κύριο Μπράιαν Σίμψον που ήταν ο σκιώδης εισηγητής. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επικοδομητικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε μια ισόρροπη συμβιβαστική λύση αποδεκτή όσον αφορά τους ε, ε, συνομοθέτες παρότι υπήρξε μια μικρή πλειοψηφία από πλευρά Συμβουλίου. Υψηλή προτεραιότητα επετέφθη στις 16 Ιουνίου σε συνάντηση των Υπουργών, όπου τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν ένα γενικό πλαίσιο προσέγγισης για την ε, ενιαία οδηγία για τους σιδηροδρόμους ε, με πλειοψηφία, ώστε να επικαιροποιηθεί και να διασφαλιστεί ένα πλαίσιο για το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο μέτρων για την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, αυτό που κάναμε ήταν διεξαγάγαμε περίπλοκες σύνθετες ε, διαπραγματεύσεις ευθυγραμμιζόμενοι προς τους στόχους της Βελγικής Προεδρίας προηγούμενα όπου, όπου υπήρχαν επιφυλάξεις ε, που είχαν διατυπωθεί σε σχέση με τους κυριότερους άξονες ε, των προτάσεων. Και σαν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από πλευράς μας καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια ισόρροπη συμβιβαστική λύση μεταξύ των κρατών μελών που είχαν διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις. Και έτσι Τούτων λεχθέντων μπορώ να πω ότι πιστεύω ότι αυτός ο συμβιβασμός θα παράσχει στις μελλοντικέ προεδρίες ε, ένα ισχυρό θεμέλιο, ένα επαρκές περιθώριο ελιγμών και ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό που θα είναι αποδεκτός και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο ήταν κύρια προτεραιότητα για την Ουγγρική Προεδρία να προαγάγουμε τις ε, ποτάμιες πλωτές μεταφορές ε, και να ε, δραχθούμε των ευκαιριών που θα παρήχονται. Δεσμευμένοι προς αυτό το στόχο διεξαγάγαμε μια συνεδρίαση υψηλού επίπεδου στο Estergom για την ένταξη των πλωτών ποτάμιων μεταφορών και τη συνεισφορά τους στην οικονομία και για την χρηματοδότηση στο μέλλον του προγράμματος ΝΑΙΑΔΕΣ. Και βασιζόμενοι στα συμπεράσματα αυτής της διάσκεψης, υιοθετήσαμε συμπεράσματα από πλευράς του Συμβουλίου στις 16 Ιουνίου 2011. Εγκρίναμε τα συμπεράσματα αυτά και σε αυτό το έγγραφο τα κράτη-μέλη ε, πρότειναν σαφείς ε, κατευθυντήρες γραμμές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συνέχιση αυτού του προγράμματος στο μέλλον. Και όσον αφορά την ε, ολοκλήρωση και την ε, ένταξη σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, η Ουγγρική Προεδρία ανέλαβε πρωτοβουλία για τον, τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς για τις ενέργειες μεταφορές. Και ήδη τον ε, Μάρτιο στη Βουδαπέστη είχαμε μία διάσκεψη το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τα, ε, τις λειτουργικές ομάδες ή κατηγορίες καθώς και η διαλειτουργικότητα των σημερινών και μελλοντικών συστημάτων και την εφαρμογή των ενιαίων εθέρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, θα πρέπει εδώ να ληφθούν υπόψη ε, τα μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα εκείνα μέτρα που είναι αναγκαία. Τέλος, εξίσου σημαντικό ένα από τα σημαντικότερα θέματα που μας ανέμενε ήταν διτού χαρακτήρα, διπλό. Έπρεπε να αξιολογήσουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση όσον αφορά τα προγράμματα Έγνος και Γαλιλαίο και έπρεπε επίσης να εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε μελλοντικές προτεραιότητες ιδιαίτερης σημασίας, ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε ένα αποτέλεσμα έντονων σε βάθος διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών ήταν βρέθηκε σε θέση να υιοθετήσει τα συμπεράσματα με πρόταση του Συμβουλίου στη συνεδρίαση του Μαρτίου, μόνο δύο μήνες μετά την δημοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα συμπεράσματά του ομόφωνα επιβεβαίωσε επαλήθευση τη δέσμευσή του υπέρ αυτών των προγραμμάτων το Συμβούλιο και παρέσχε κατευθυντήρες γραμμές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προπαρασκευή νομοθετικού έργου για την κατάρτιση και χρηματοδότηση μετά το 2013 προτεραιοτήτων και δράσεων. Και τώρα όσον αφορά στη συνέχεια τις διοργανικές διαπραγματεύσεις για το σχέδιο απόφασης όσον αφορά τους κανόνες προσπέλασης, προσβασιμότητας για τις δράσεις Γαλιλαίου. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες και σε βάθος με επιτυχία ολοκληρώθηκαν υπό την Ουγγρική Προεδρία κατά την πρώτη ανάγνωση κιόλας, στην φάση της πρώτης ανάγνωσης. Όσον αφορά την ασφάλεια και συνολικά τα θέματα ασφάλειας, θα ήθελα να αναφέρω τη διαπραγματεύσεις για το σχέδιο οδηγίας για την διευκόλυνση της ανταλλαγής διασυνοριακά στοιχείων που αφορούν παραπτώματα, παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τη δίωξη των παραβατών, οι διαπραγματεύσει λίμναζαν από το 2008. Αυτή η οδηγία για τη δίωξη παραβάσεων του ΚΟΚ, ε, κώδικα οδική κυκλοφορία έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή των πολιτών και μπορούν να συνεισφέρουν υπέρ της οδική ασφάλειας. Σαν αποτέλεσμα έντονων τριμερών διαλόγων από πλευράς μας ήταν δυνατόν με επιτυχία να ολοκληρωθούν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις σε δεύτερη ανάγνωση υπό την Ουγγρική Προεδρία και να ευστευτεί ε, με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά την ολομέλειά του στις 6 Ιουλίου στο Στρασβούργο αυτές τις προτάσεις και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο έδρασαν με ιδιαίτερη ευθύνη, με ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Με αυτή την απόφαση αποδείχθηκε ότι συνεργαζόμενοι προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών είμαστε πραγματικά σε θέση να επιτύχουμε σημαντικέ βελτιώσει. Ιδιαίτερε ευχαριστίε στοχεύουν προ την κυρία Γιάλα Σέντερ, η συγγήτρια του Ευρωκοινοβουλίου, για το επικοδομητικό πνεύμα που κατέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Άλλα χαρτοφυλάκια στον τομέα της ασφάλειας είναι τα χαρτοφυλάκια, δύο χαρτοφυλάκια για τις ε, ε, μεταφορές. Η Ουγγρική Προεδρία βασίστηκε στην υποστήριξη του εταίρου του Βελγίου στην Τρόικα των Προεδριών, πράγμα το οποίο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο η υπουργική συζήτηση για την τροποποίηση των ε, τρεχουσών διαδικασιών όσον αφορά την υπηρεσία ε, θαλάσσιων ε, πλωτών μεταφορών εγκρίθηκε κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών. Με βάση αυτή την απόφαση καταφέραμε να επιλύσουμε τα θέματα που εκκρεμούσαν και υιοθέτησε μια γενική προσέγγιση για αυτή την πρόταση το Συμβούλιο στη συνεδρίασή του κατά τις 16 Ιουνίου 2011. Και έτσι επίσης καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία επί του κειμένου για το κείμενο της απόφασης ε, για την Ευρωπαϊκή την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο της ε, Σύμβασης των Αθηνών του 1974 που είναι η σύμβαση που αφορά τα δικαιώματα επιβατών και της μεταφοράς επιβατών και αποσκευών διαθαλάσσης. Όσον αφορά την ασφάλεια, όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές θα ήθελα σχετικά να αναφερθώ σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο όπου επετεύχθη συμφωνία πάλι υπό την Ουγγρική Προεδρία κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά την 31η Μαρτίου. Απόφαση του Συμβουλίου ελήφθη για την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Διεθνούς ε, Ένωσης ε, Πολιτικής Αεροπορίας, ΙΚΑΟ. Με βάση αυτά υπέγραψαν οι εταίροι τα συμβαλώμανα μέρη την, το πλαίσιο συμφωνίας και υιοθέτησαν, ενέκριναν και το πρώτο παράτημα για την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών. Κάνοντας λόγο για την ασφάλεια στις εναέριες μεταφορές, θα ήθελα φυσικά να αναφερθώ και στην έκρηξη του ηφαιστείου Γκρίμσβατον στην ε, Ισλανδία που ε, δημιούργησε προβλήματα και την θέσπιση της ε, ζώνης ε, απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την ε, Ισλανδία αποφασίσαμε και με, από κοινού με τον Αντιπρόεδρο Κάλλας τα μέτρα που έπρεπε να υιοθετηθούν. Νέες διαδικασίες, νέες διεργασίες απέρευσαν από τα όσα συνέβησαν πέρυσι. Με βάση αυτές τις διεργασίες κατάφεραν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά την κατάσταση. Εν τέλει, θα ήθελα να πω λόγια για άλλα χαρτοφυλάκια για τις διεθνείς μεταφορές που δεν ανέφερα μέχρι τώρα αλλά που και αυτά τα διαπραγματευτήκαμε κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας μας. Απόφαση ελήφθη για την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμβαση της ε, μεταφοράς ε, σιδηροδρομικά και για την ε, ε, σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΤΙΦ, ε, την Διεθνή Οργάνωση όσον αφορά τις ιδεοδρομικές μεταφορές. Η συμφωνία υπεγράφει κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΤΙΦ στο, στην Βέρνη διεθνείς διαπραγματεύσεις ήταν εξίσου σημαντικές υποθέσεις για την Ουγγρική Προεδρία. Σαν συνέπεια τούτου κάναμε τα εξή. Διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν με την Μολδαβία για μια σφαιρική συνολική συμφωνία για τις ενέργειες μεταφορές. Επίσης ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την πιθανή συμπερίληψη των δικαιωμάτων μικρής ακτοπλοείας, ε, ε, μικρών διαδρομών, καμποτάζ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Ελβετία. Μια ευρεία συμφωνία για τις μεταφορές υπεγράφει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας. Ισλανδία και Νορβηγία προσχώρησαν στην σφαιρική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ που τροποποιήθηκε με ένα πρωτόκολλο που προσαρτήθηκε σε αυτήν. Η Ουγγρική Προεδρία επίσης πέτυχε σημαντικές επιτυχίες στην διεθνή συνεργασία όσον αφορά την δορυφορική ναυσιπλοεία και δορυφορική ναυτιλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εντολή από πλευράς του Συμβουλίου να ολοκληρώσει, να προβεί σε ολοκλήρωση σε συμφωνίες ε, για την ε, έναρξη και ολοκλήρωση των συμφωνιών με τη Χιλή και τη Βραζιλία. Ζητήσαμε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συναφή θέματα, για συμφωνία δορυφορικής ναυτιλίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Συνάψαμε επίσης συμφωνίες ε, για την προώθηση διατάξεων και την χρήση του Γαλιλαίου και της ε, δυνατότητας έβρεσης ε, γεωγραφικού στίγματος μέσω των, της δορυφορικής ναυσιπλοείας και των δυνατοτήτων του Γαλιλαίου. Με ικανοποίηση μπορώ να σας αναφέρω ότι η Ουγγρική Προεδρία κατάφερε να έχει θετικά αποτελέσματα και να επιτελέσει θετικό έργο όσον αφορά τις δεσμεύσεις που είχε υπομειστεί, που είχε αναλάβει για θέματα μεταφορών. Επιτρέψτε μου συντομία να αναφέρω και την ε, στρατηγική για τη λεκάνη του Δούναβη, όπου αποφάσεις υιοθετήθηκαν στις 24 Ιουνίου 2011 αυτή η στρατηγική είναι η δεύτερη πρωτοβουλία, η δεύτερη σε σχέση με την διαπεριφερειακή στρατηγική που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμονίζοντας τις διασυνοριακές διατάξεις και διεργασίες για 14 κράτη-μέλη που αφορώνται από το Δούναβι. Οκτώ κράτη-μέλη βρίσκονται ε, εντό και έξι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η στρατηγική υποστηρίζει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και μπορεί να συνεισφέρει στο να είναι βιώσιμη και να προαχθεί η αηφορία στην λεκάνη του Δούναβη, συνεισφέροντας την ανάπτυξη προγραμμάτων και σχεδίων που θα υλοποιούνται και θα εφαρμόζονται από τους εταίρους, από τα συμβαλόμενα μέρη. Αυτή η στρατηγική έχει δύο συνιστώσεις, δύο άξονες που αφορούν τις μεταφορές. Ανάπτυξη της κινητικότητας σαν αποτέλεσμα επενδύσεων στις υποδομές, ιδιαίτερα στον άξονα μεταξύ διασύνδεσης βορρά και νότου. Και δεύτερον, την προώθηση των πλωτών ε, ποτάμιων μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τις φιλοπεριβαλλοντικές πτυχές και πολιτικές. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω ότι αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν μόνο να επιτευχθούν με βάσει την στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που ήταν αναγκαία προϋπόθεση της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ημών του Ευρωκοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και εκφράζω τις ευχαριστίες από πλευρά της, της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου, της Ουγγρικής Προεδρίας ε, για αυτή τη στάση. Το έργο μας νομίζω ότι μπόρεσε να αποδείξει την δέσμευση της Ουγγαρίας και την ευδοκίμηση των στόχων για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Επίσης ε, εκφράζω την ελπίδα ότι με βάση αυτή τη δουλειά μας συνεισφέραμε στην θέσπιση και δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές που θα εξυπηρετεί τη δημιουργία και προώθηση μιας πιο ενωμένης, ολοκληρωμένης, πιο ανταγωνιστικής και πιο φιλοκοινωνικής Ευρώπης που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο μέλλον. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προβλέπω στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την επισκόπηση της ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Ο κύριος Γκρός, η κυρία Γέλα Σέντερ και ο κύριος Κόζα έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Γκρός λοιπόν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ εξ ονόματο της ομάδας μας θέλω να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία. Η Προεδρία σας ήταν μια πολύ δραστήρια Προεδρία. Δεν ανήκε στι Προεδρίες που δεν κατάφεραν να πετύχουν πολλά, πολλά παρά μόνο τα εύκολα, ε, τους εύκολους καρπούς ε, μπόρεσαν να δρέψουν. Εσείς καταβάλατε προσπάθειες ε, που ήταν δύσκολο, δυσχερές εγχείρημα και δρέψατε καρπούς που ήταν σημαντικοί. Ήταν σημαντικό όχι μόνο για τα σημαντικά χαρτοφυλάκια ότι τοποθετηθήκατε και δώσατε μια πρώτη τοποθέτηση για το λευκό βιβλίο, αλλά και για τις διασυνοριακές ανταλλαγές και ε, διάχυση στοιχείων και πληροφοριών, αλλά είναι σημαντικό ότι κινητοποιήσατε το Συμβούλιο να καταλήξει σε απόφαση. Για παράδειγμα, στα ΦΑΠΣ είχατε μια πολύ σημαντική διάσκεψη το Μάρτιο και ο συντονιστής μας κύριος Γιαζεμπόφσκι με ικανοποίηση το είδε αυτό διότι δώσατε χαρακτηριστικά και κατευθύνσεις ως χώρα στις 5 Μαΐου είχατε την κρατική σύμβαση που υπεγράφει σε σχέση με αυτό το κέρια σημασία θέμα για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών. Ήταν ένα εξαιρετικό επίτευγμα έπρεπε να πιστούν και εκείνοι που έπρεπε να υπογράψουν και με το καλό παράδειγμα που δόθηκε αυτό νομίζω ήταν θετικό για τους υπόλοιπους και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνατε. Φυσικά το ότι δεν είμαστε πάντα όλοι ικανοποιημένοι με όλα τα επιτεύγματα ή αποτελέσματα του Συμβουλίου, το γνωρίζετε αυτό. Πρόκειται για συμβιβασμό που επετεύθηκε η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και από πλευρά εισηγητού σε αυτά τα δύο χαρτοφυλάκια για την Ευρωβινιέτα για παράδειγμα για, τις, ε, ε, για τα θέματα οδικών μεταφορών υπήρξε πολύ, πολύ αυθεντικά παραγωγική δουλειά. Ελπίζω ότι από το Συμβούλιο το ίδιο θα καταδειχθεί περισσότερο φιλευρωπαϊκή νοοτροπία και δράση διότι πιστεύουμε ότι οι εθνικές, τα εθνικά συμφέροντα σε αυτόν τον τομέα δεν εξυπηρετούν καθόλου την Ευρώπη και πρέπει να προχωρήσουμε πιο φιλοευρωπαϊκά. Θα ήθελα για δύο θέματα να έχω την αξιολόγηση και τοποθέτησή σας. Πρώτον, είχαμε προηγούμενα συζήτηση για τους αρωτές σώματος στον τομέα ανείχνευσης στα ε, υγρών και ουσιών στα αεροδρόμια και είπαμε ότι μέχρι το 2013 πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προπαρασκευασμένοι. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναβιώσουμε αυτά τα οποία βιώσαμε φέτος. Δηλαδή μόνο μία βραχυπρόθεσμη απάντηση εφήμερα των κρατών μελών που απεμπολούν εκείνα τα οποία έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευτεί τα ίδια τα κράτη-μέλη να επιτελέσουν. Πώς βλέπετε εσείς αυτόν τον τομέα για το μέλλον στη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, διότι αυτά τα οποία μονομερώς ας το πούμε έτσι συνέβησαν και σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν καλό παράδειγμα και ελπίζουμε δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Δεύτερον, υπήρχαν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Εγώ πιστεύω ότι το μέλλον σε αυτό το χαρτοφυλάκιο θα εξαρτηθεί από το θάρρος των κρατών μελών να μειώσουν τον αριθμό των προγραμμάτων αυτών και να υπάρξει πιστικό έργο σε κυριότερους άξονες που θα δημιουργηθούν. Πώς το αξιολογείτε εσείς αυτό. Και ίσως εδώ ένα τελευταίο σημείο στο οποίο δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτά τα οποία ελήφθησαν ως αποφάσει. οι προτάσεις έγιναν από το Συμβούλιο για το σιδηρόδρομο, για τους σιδηροδρόμους. Δεν είναι μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη προσέγγιση για τους σιδηροδρόμους. Εδώ εξακολουθούν και υφίστανται εθνικές απόψεις ή συμφέροντα σε πολλούς τομείς. Σε σχέση με την Ουγγρική Προεδρία, Πιστεύω ότι με κάποια κράτη θα πρέπει να σταματήσει αυτή η τάση αν θα έχει ε, προοπτική για το μέλλον ε, η δράση στους σιδηροδρόμους, μόνο ευρωπαϊκή θα είναι αυτή η προοπτική. Και οι σιδηρόδρομοι ως πλήρης ισότιμος εταίρος των άλλων μεταφορών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχετε την εντύπωση ότι μπορούν, μπορούν οι σιδηρόδρομοι να βρεθούν σε καλύτερη πορεία με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στο μέλλον. Ευχαριστώ. κυρία Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω ότι ο κύριος Σάιτερ Χαντράου, ο συντονιστής μας, ήθελε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς ε, είχε ένα πρόβλημα, είχε μια λυμένη υποχρέωση και δεν μπόρεσε να έρθει. Και λυπάται που δεν μπορεί να σχολιάσει και ο ίδιος τα αποτελέσματα της Ουγγρικής Προεδρίας. Είδαμε τελικά την ιδέα αυτή της Τρόικας. Δρομολογούν οι προηγούμενες προεδρίες κάποια θέματα, αλλά τελικά η, κάθε φορά η εκάστοτε προεδρία είναι αυτή η οποία ε, βάζει τους στόχους και ολοκληρώνει κάποια πράγματα. Και στους τομείς που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας, ε, η Προεδρία σας έχει καταφέρει να κλείσει, να ολοκληρώσει πολύπλοκα θέματα, κάποια παλαιότερα ή κάποια πολύ επίχημαχα. Κατάφερε λοιπόν να τα ολοκληρώσει με στένος, ε, με όθηση και κάποιες φορές ε, κινδυνεύοντας. Γιατί οι νέες προεδρίες έχουν πολλές φορές αυτή την όθηση, αυτή την όρμη. Καταφέρατε λοιπόν να κλείσετε κάποια θέματα. Και νομίζω ότι υπάρχουν πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία για τις επόμενες προεδρίες και τα τελευταία που είπατε. Βέβαια το πιο πολύπλοκο θέμα, του οποίου είχαμε ένα αποτέλεσμα, που νομίζουμε ότι είναι αρκετά σημαντικό, είναι το θέμα της Ευρωβινιέτας 3,5 για τον κύριο Χαντράου. Νομίζω ότι λόγω της επιμονής του κ. Χαντράουι και της ε, διαπραγματευτικής του ικανότητας καταφέραμε μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να καταλήξουμε σε συμφωνία επί αρχών πολύ σημαντικών όπως ε, παραδείγματος χάρη ο Ιππένον πληρώνει. Αυτό πλέον εγγράφεται στην πολιτική των οδικών μεταφόρων παρά τις πολλές ε, αντιστάσεις. Επίσης άλλες πτυχές σε ό,τι αφορά τα έσοδα και τη μεγαλύτερη διαφάνεια της εσωτερήκευσης του εξωτερικού κόστους. Επίσης σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος που θα προετοιμάσει μελλοντικές εφαρμογές. Μια σημαντική προστιθέμενη αξία είναι ότι ξεκίνησε ο εθνικός διάλογος ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την ε, απόδοση κάποιων εισόδων, για, δηλαδή σηματοδοτούνται κάποια ποσά για συγκεκριμένους ε, στόχους. Και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το 15% το οποίο θα πρέπει να προβλέπεται για τα ε, δίκτυα, τα διευρωπαϊκά. Και επίσης ε, τα ιδιαίτερος χαρακτήρες των ορεινών περιοχών που ελήφθη υπόψη. και θα πρέπει επίσης από το 2015 να έχουμε το Euro 3 ε, και ανανέωση του στόλου. Έχουν ε, τεθεί τα θεμέλια, δεδομένης και της κρίσης δεν ήταν εύκολα να επιτευχθεί πρόοδος, αλλά νομίζω ότι έχουμε παρόλα αυτά καταφέρει αρκετά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, ελπίζω σε σχέση με τη χρηματοδότηση κυρίως, να είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Η πρώτη πρόταση της Κομισιόν στον τομέα των μεταφορών, στο πλαίσιο ενός δημοσιονομικού πλαισίου, που δεν είχε να κάνει βέβαια με την αναθεώρηση των δικτύων, αλλά τις δημοσιονομικές προοπτικές, ξέρετε ότι ε, είχε ως αποτέλεσμα αντιδράσει στη χώρα μου, στην Ιταλία κτλ. Περίπλοκα είναι τα πράγματα λίγο. Και ελπίζω και τα συμπεράσματά σας να βοηθήσουν στην ε, λήψη καλύτερων αποφάσεων ε, στο μέλλον στο Συμβούλιο. Πάντως θέλω να σας συγχαρώ για τα συμπεράσματα σας και σε ό,τι αφορά ε, ε, την ποτάμια ε, και το πρόγραμμα Ναϊάδες που είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να συνεχιστεί και που είναι λίγο τώρα μετέωρο. Και ότι καώ δεν είναι εδώ, αλλά είμαι βέβαιη ότι και η ίδια θα σας συγχαρεί σε ό,τι αφορά την όθηση της στρατηγική για το Δούναβη. Ήταν κάτι πολύ αναγκαίο να βελτιωθεί η ποτάμια ε, ναυσιπλοεία. Και δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, γι' αυτό ολοκληρώνω με, τις διασυνοριακά, με τα διασυνοριακά πρόστιμα. Ήδη με τη Βελική Προεδρία είχαμε ξεκινήσει. Ίσως να μην είναι ε, θέμα που έχει να κάνει με τις μεταφορές. Ψάχνουμε να το βρούμε ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνη. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Για μα έχει να κάνει με τι μεταφορέ, Έχουμε τη ρητραναθεώρηση εν μέρη και μπορούμε να επανέλθουμε σε μια βάση και τις μεταφορές τη επόμενη διαπραγματεύσεις. Να σας ευχαριστήσω πάντως θερμά γιατί πράγματι η Βελγική Προεδρία είχε ήδη προετοιμάσει αυτό το πακέτο αλλά έμενε ένα θεμελιώδες κομμάτι που ήταν αυτό της προσαρμογής του συστήματος Εουκάρης έπρεπε να γίνει προσαρμογή. Ήταν πολύπλοκο εγχείρημα, γιατί υπήρχαν τα ζητήματα προστασίας δεδομένων, ανταλλαγής, χρήσης δεδομένων και βέβαια με το χειρό των κρατών μελών. Και θέλω να σας συγχαρώ γιατί πραγματικά επιδείξατε ικανότητα και μεγάλη γνώση και εμπειρία για να έχουμε αυτή την προσαρμογή. Στι διαπραγματεύσει που είχαμε ήσασταν ιδιαίτερα επιδεκτικοί απέναντι στι θεμητέ ανησυχίε των Ευρωβουλευτών για την ανάγκη αύξηση τη προστασία των δεδομένων, την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, τον έλεγχο αυτών των δεδομένων από τον ενδιαφερόμενο και μας διαβεβαιώσατε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιμόλυνση με οποιοδήποτε άλλο φάκελο ή οποιοδήποτε άλλο τομέα πέραν της οδηγίας, πέραν του παιδί εφαρμογής της Το θέμα επίσης ε, της κοινοποίηση και της ε, λήψης της κοινοποίηση και το σχετικό με τις οικογένειες των θυμάτων ε, των τροχαίων. Γενικά νομίζω ότι καταφέραμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Εκεί που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα διευκόλυνε τη συνένεση για τους πίνακες συσχέτισης που είναι ένα διοργανικό με βέβαια θέμα και του οποίου μένεται ακόμα η μάχη στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, καταφέρατε να σημειώσετε κάποια πρόοδο σε σχέση με αυτό το οποίο έγινε με την Ευρωβινιέτα, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Εμείς υπήρξαμε γεννόδοροι ως Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι εσείς θα μπορούσατε να είχατε βοηθήσει να σημειωθεί πρόοδος και σε επίπεδο ε, Συμβουλίου. Επειδή θα κοπανίσει το σφυρί ο πρόεδρος όπου να είναι, Νομίζω ότι ε, πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ε, για, για τα πρόσφατα που σας είπατε μπορούμε να έχουμε και έτσι ένα κοκτέιλ για να το γιορτάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σχεδίαζα να παρέμβω για μεγαλύτερο διάστημα, αλλά οι προλαλήσαντες έθεσαν ακριβώς τα ερωτήματα που ήθελα εγώ να διατυπώσω. Μία και μόνη ερώτηση απομένει που ήθελα να διατυπώσω. Πρωτού όμως διατυπώσω αυτή την ερώτηση θα ήθελα να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία παρακολούθησα την πρόοδο που επετελέστη και το έργο που ολοκληρώθηκε και μπορώ ειλικρινά νομίζω να πω και νομίζω την ομόφωνη απόφαση στον τομέα των πολιτικών μεταφορών η Ουγγρική Προεδρία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, κατάφερε όλους τους στόχους της να τους επιτελέσει. Ένα θέμα το οποίο απομένει είναι το δικαίωμα επιβατών. Για μένα σημαντικό θέμα. Ποια είναι η πρόοδος η οποία επετεύχθη στα δικαιώματα επιβατών στις μεταφορές. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Και τέλος, να πω και εγώ από πλευράς μου κάποια πράγματα. Να επαναλάβω τις απόψεις ε, που εξέφρασαν και κάποια άλλα μέλη για την Ουγγρική Προεδρία. Νομίζω ότι η Ουγγρική Προεδρία επέτυχε πολλά. Σαφώς ε, κατάφερε να προωθήσει δύο μεγάλα ζητήματα, αλλά ε, νομίζω και τα όσα έκαναν σε άλλους τομείς αξίζουν συγχαρητηρίων ξεκίνησαν κάποια προγράμματα, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα του Δούναβη. Η Επιτροπή μας ερωτεύτηκε το Δούναβη, σχεδόν τον υιοθετήσαμε, κυρίως γιατί η κυρία Τσικάου δεν μας αφήνει ποτέ να τον ξεχάσουμε το Δούναβη. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ποταμό, ο οποίος ε, υποχρησιμοποιείται και έχει τεράστιες δυνατότητες εκμετάλλευσης. Εκτιμώ ιδιαίτερα λοιπόν την Ουγγρική Προεδρία, ιδίω για τα όσα έκανε σε θέματα μεταφορών και ευχαριστώ και εσά προσωπικώ, αλλά και το προσωπικό σας ε, και τη μόνιμη αντιπροσωπεία σας διότι έκαναν πολύ σκληρή δουλειά ώστε η προοδή αυτή να οδηγηθεί στο επιτυχές αποτέλεσμα στο οποίο ε, οδηγήθηκε. Έχουμε ακόμα προβλήματα, έχουμε τους πίνακες αντιστοιχίας που είναι ε, θέμα συντονισμού. Δεν μπορούμε να σας κατηγορήσουμε ότι δεν κάνατε τίποτα βέβαια από αυτού, διότι είναι θέμα ανωτέρων ε, ευφυών ε, από ότι μας. Μας αν, απογοητεύει λίγο ότι έχει σταματήσει το θέμα των των προστήμων. Ελπίζω να τα προχωρήσει η Πολωνική Προεδρία. Και επίσης νομίζω ότι μία από τις πολύ σημαντικέ παρακαταθήκες που αφήνεται ω Προεδρία είναι το γεγονός ότι καταφέρατε να κάνετε κάποια πράγματα όταν εμείς θεωρούσαμε ότι η σχέση μεταξύ Συμβουλίου Συμβουλίου Υπουργών και του Κοινοβουλίου ήταν στο κατώτερο δυνατό επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό δεν είναι επίκριση προς την Ουγγρική Προεδρία. Στην πράξη είναι συγχαρητήρια διότι καταφέραμε να επιτύχουμε τόσα πολλά όταν στην πραγματικότητα η εμπιστοσύνη μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών και του Συμβουλίου Υπουργών ε, ήταν χαμένη υπόθεση. και μάλιστα κορυφώθηκε αυτή η αποτυχία στα όσα είχαμε τον Απρίλιο με τα υγρά και τα, τις γέλες και τα θέματα ασφαλείας. Ο κύριος Γκρός νομίζω ότι το ανέφερε. Καταφέραμε να ε, συνεργαστούμε μαζί σας, ε, διότι εσείς ήσασταν αυτούς που πήγατε στο Υπουργικό Συμβούλιο και δώσετε το παράδειγμα για το πώς πρέπει να συνεργαζόμαστε. Ε, όλοι παναχώρησαν πίσω από τα εθνικά του σύνορα για όλες τις μορφές μεταφορών και αυτό είναι κρίμα γιατί τα ευρωπαϊκά ιδανικά δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς. Το είδαμε άλλωστε και η διεισόμαση στο άτυπο συμβούλιο στη Βουδαπέστη όταν συζητούσαμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δώσουν προτεραιότητα στα διευρωπαϊκά δίκτυα και όλα τα κράτη-μέλη ήταν πρόθυμα υπό την προϋπόθεση τα δικά τους τα σχέδια να μην διαγραφούν από τις καταλόγους. Θα σας χρησιμοποιούμε λοιπόν στο μέλλον ως ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου Υπουργών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως την Προεδρία σας μία από τις πιο επιτυχείς Προεδρίες σε συνέχεια μάλιστα και της Βελγικής Προεδρίας που ήταν αρκετά καλή. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που θα θέσουμε στο συνάδελφο από την Πολωνία ε, σήμερα το απόγευμα ε, είναι κατά πόσο θα θελήσει να έχει μια τρίτη επιτυχή Προεδρία στη σειρά. Ε, κύριε Υπουργέ, να σας δώσω το λόγο όμως για να απαντήσετε κάποια από τα θέματα που ετέθησαν εδώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσω με την οδηγία για την Ευρωβινιέτα. Όλοι γνωρίζουμε φυσικά ότι κατά τα έλλη του, τέλη του 2010 ολοκλήρωσε αυτό το χαρτοφυλάκιο η Βελγική Προεδρία και έτσι καταφέραμε, μπορούσαμε να το υποβάλουμε ως πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα ε, επετεύθη η αναγκαία πλειοψηφία στο Συμβούλιο σαν δεν είχε επιτευχθεί ακόμα η πλειοψηφία στο Συμβούλιο, υπήρχαν κάποια προβλήματα και όταν ήρθα να συναντήσω το Κοινοβούλιο ανέφερε ότι βασιζόμαστε στην ελαστικότητα και στην δική σας θετική στάση διότι δεν υπήρχε περιθώριο λιγμών στο Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν μπόρεσε να στεφθεί με επιτυχία μετά από αυτή την ε, τοποθέτηση. Χρειαζόταν η βοήθεια του Κοινοβουλίου για να στεφθεί με επιτυχία η πρωτοβουλία της Ουγγρικής Προεδρίας διότι διαφορετικά δεν θα είχαν υιοθετηθεί οι συμβαστικές μας προτάσεις από το Συμβούλιο και δεν θα είχε στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων στο Συμβούλιο υπήρχαν υπουργοί που έπρεπε να τους καλέσω τηλεφωνικά και να συζητήσω τα εκκρεμούντα θέματα μαζί τους ε, για να, μπορέσω να, κατα... να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισχνή πλειοψηφία και να καταλήξουμε στο ε, Ευρωκοινοβούλιο με την πρότασή μας και στη συνέχεια έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτό το χατοφυλάκι. Ομολογώ ότι δεν καταφέραμε σημαντική πρόοδο. Δεν ήταν ένα γιγάντιο άλμα προς τα εμπρός. Όμως ε, βασιζόμαστε σε αυτή την πολιτική βάση. Ελπίζω ότι θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα εξίσου και όσον αφορά την ασφάλεια και θέματα ασφάλειας στα αεροδρόμια θα πρέπει να πω ότι ναι, στις 9 Απριλίου 2000, η συμφωνία δεν είχε επιτευχθεί. Βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαστε μόνο εμεί ε, που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Α δούμε τι ΣΥΠΑ και την προσέγγιση που υιοθετούν οι ΗΠΑ. Υπάρχουν εδώ οι διεθνεί ε, παράμετροι που δεν μπορούμε εμεί να επηρεάσουμε και όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συνεξετάζονται. Και φυσικά τα θέματα ασφάλεια πρέπει να είναι ύψη τη προτεραιότητα πάντα και δεν πρέπει βιαστικά να αντιμετωπίζονται, διότι μπορεί ύστερα να καταλήξουμε, αν είμαστε υπερβολικά να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την η ασφάλεια. Όσον αφορά την χρηματοδότηση, υπήρξε μια συνάντηση των Υπουργών στο Γκέντελε, όπου είχε ε, εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα της χρηματοδότησης. Και πιστεύω ότι ένας συμβιβασμός βρίσκεται υπό εξέλιξη η χρηματοδότηση πιθανότατα θα αυξηθεί η συγχρηματοδότηση. Το επίπεδο χρηματοδότησης όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα είναι υψηλότερο τελικά, αλλά ταυτόχρονα αυτό που πετύχαμε είναι να εγκριθεί μια άλλη πρόταση, άλλα κράτη-μέλη τα οποία θα είναι επιλέξιμα για διαθροτικές τέτοιες δράσεις και θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμα για την ε, χρηματοδότηση, για κονδύλια, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα καθώς επίσης και για την προώθηση των υποδομών. Τα σχόλιά σας είναι δικαιολογημένα. Ο λόγος για τον οποίο δεν καταφέραμε να πετύχουμε μια πρόοδο είναι η χρηματοοικονομική κρίση, οι πρόσφατες εξελίξεις. Δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει αυτή την κρίση και πρέπει να δεχθούμε ότι η πρώτη και κύρια προτεραιότητα θα είναι η οικονομική σταθερότητα και σταθεροποίηση. Όμως ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτούς τους στόχους. Τώρα, για το πακέτο για τα μέτρα για τους σιδηροδρόμους επισκοπώντας και βλέποντας το τι συνέβη με την ιστορία για, ε, για αυτό το πακέτο, πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Γκρός ποτέ δεν επιτυγχάνονται σημαντικές πρόοδοι σε μικρή χρονική περίοδο, σε μικρό χρονικό διάστημα. Όμως καταφέραμε να επιτύχουμε μια κάποια συγκεκριμένη πρόοδο και αυτό το θεωρώ σημαντικό. Το ίδιο ισχύει και για την οδηγία για την Ευρωβινιέτα, διότι η Βελγική Προεδρία ολοκλήρωσε το δικό της μέρος σε αυτό το έργο. Κατανοώ ότι το περιθώριο λιγμών ήταν περιορισμένο, όμως τουλάχιστον τώρα έχουμε ένα κάπως μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών και Πολωνική Προεδρία που ακολουθεί την δική μας είναι και αυτή από ό,τι φαίνεται πολύ φιλόδοξη και έτσι εξακολουθώ να ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα ευδοκιμήσουν αυτές οι ελπίδες και από πλευράς των κρατών μελών που προσπαθούν να ε, παρουσιάσουν και να διαφυλάξουν τα δικά τους συμφέροντα. Και είναι δύσκολο πολλές φορές να τύχουν ιδιαίτερης προτεραιότητας οι ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες. Πρέπει με μικρά βήματα να προχωρήσουμε, να είμαστε υπομονετικοί, να δείξουμε καρτερία και ανθεκτικότητα για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο βήμα προς βήμα. Και μετά η χρήση κονδυλίων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημιουργία αυτού του συστήματος. Ένας συμβιβασμός νομίζω επετεύχθη. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν ένα σχετικά μεγάλο περιθώριο ελιγμών όσον αφορά την υλοποίηση και χρήση των κονδυλίων αυτών. Όμως είναι προφανές, είναι πρόδειλο ότι οι υποδομές, για τα θέματα των υποδομών υπάρχει πάντα μεγάλη ανάγκη, υπάρχει δίψα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ε, και να διατεθούν τα αναγκαία χρήματα και αν μπορούν αυτά τα πράγματα να ε, προαχθούν τότε θα ήταν ικανοποιημένο και το Ευρωκοινοβούλιο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι ε, ποτάμιες πρωτές μεταφορές και η πολιτική για τον Δούναβη. Πραγματικά ελπίζω ότι η συνέχιση του προγράμματος Ναϊάδες θα μπορέσει να συνεχιστεί και μετά το 2013, διότι επιπρόσθετα πέρα από τους σιδηροδρόμους και αυτό είναι ένας τομέας φιλοπεριβαλλοντικών μεταφορών και αυτό είχε εκτεθεί και είχε τονιστεί στο Λευκό Βιβλίο και έτσι με αυτή την πολιτική των πλωτών ε, ποτάμιων μεταφορών μπορούμε φιλοπεριβαλλοντικά να επιτύχουμε τους φιλοπεριβαλλοντικούς μας στόχους και για τη διάχυση πληροφοριών και ε, την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά παρα... τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ένα θέμα πολυσχηδές που καλύπτει πολλές παραμέτρους αφορά την, τα ιδιωτικά δεδομένα της προσωπικής ζωής, τα στοιχεία ε, των παραβατών. Πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν με τον, ε, έπρεπε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο για να ευδοκιμήσει ο στόχος. Αν πραγματικά δούμε όλες λοιπόν τις πτυχές μπορούμε να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβίβασμα, ικανοποιητικό συμβίβασμα. Αναφέρθηκαν και οι πίνακες αντιστοίχησης ή σύγκριση. Νομίζω αυτό θα είναι ένα θέμα για την επόμενη Τρόικα. Εξετάζοντας το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους σχεδιάζουν και οι Πολωνοί να δώσουν συνέχεια σε αυτό και ελπίζουμε ότι θα στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα στο μέλλον. Για τα δικαιώματα των επιβατών. Ρώτησε ο κύριος Κόσα το έθεσε ερώτημα για το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι υπήρχε μια ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή αποζημιώσεων για την προστασία θυμάτων. Αυτό εισήχθη στην ομάδα εργασίας ως πρόταση στις 2 Μαΐου 2011 συζητήθηκε από τα κράτη-μέλη και με βάση αυτές τις συζητήσεις θα έλεγα ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν συμπεράσματα από πλευράς του Συμβουλίου και να προαχθεί νομοθετικό έργο. Αναμένουμε νομοθετικές προτάσεις ε, να ακολουθήσουν το 2012. Ελπίζω να μην αμέλησα κάποιο ερώτημα και να μην το ξέχασα. Όχι, όχι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Υπουργέ, θερμότατα, να επαναλάβω τις ευχαριστίες και σε σας προσωπικά και στο προσωπικό σας και στη με την προσωπία. Σίγουρα τώρα προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την Πολωνική Προεδρία. Ελπίζω ωστόσο ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις ε, σχέσεις ε, που αναπτύξαμε επί δική σας Προεδρία. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ξανασυνεργαστούμε ίσως και με διαφορετική ιδιότητα. ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται εδώ η πρωινή μας ε, συνεδρίαση. Επαναρχόμαστε στις 3 που θα έχουμε τον Πολωνό Υπουργό Μεταφορών και τον Πολωνό Υπουργό Τουρισμού μετά. Θέλετε κάτι να πείτε. Πείτε το. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω απλά ότι ελπίζω ότι έχουμε αυτό που είπα προετοιμάσει έτσι μια μικρή δεξίσωνη κοκτέιλ ε, για να πιούμε ένα ποτό με τη Γραμματεία, του Συμβουλίου, της Προεδρίας, της Επιτροπής, με όλους τέλος πάντων και για να ευχαριστήσουμε έτσι όσους μας βοήθησαν να ε, καταλήξουμε σε αίσιο πέρασμα το θέμα της ε, οδικής ασφάλειας που ήταν τόσο σημαντικό. Λοιπόν, δωρεάν ποτό έξω όποιο θέλει για το διασυνορικό έργο το οποίο έγινε επί Ουγγρικής Προεδρίας. Τρεις και πάλι και οι συντονιστές και το η γραμματεία συγκεκριμένα, να παρακαλέσω να προσελκύσει μέλη εδώ, να έρθουν βουλευτές, γιατί θα έρθει η Πολωνική Προεδρία.